Σας ευχαριστώ. Με ηρεμία να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ για την συνεργασία. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 78 εφόσον λέτε ότι δύο ταυτόχρονα αφαίρεσαν την κάρτα τους. Αρχίζει η ψηφοφορία. Παραμένει ένας υπεράριθμος. Ο ένας από το ΕΛΚ να βγάλει την κάρτα του. Πέρασε. και απερίφθη με ισοψηφία. Όντω είχαν, από ό,τι φαίνεται, βγάλει την κάρτα του ταυτόχρονα δύο συνάδελφοι του ΕΛΚ. Έτσι λοιπόν έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια. Και πάμε στην 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 81 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 84 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Αιτιολογικές σκέψεις, αιτιολογικές γνώμες, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 2 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 3 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 4 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 5 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 10 υπέρ κατά αποχές απερίφθη Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές. Α, εγκρίνεται. Ναι, ναι. Ναι, εγκρίνεται επιτέλους. Ε, καταπίπτουν οι 11 και 13 και πάμε στη 12. Υπέρ, κατά αποχές. Απερίφθη, 14 υπέρ, κατά αποχές. Απερίφθη, 15 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 16 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 17 Επαληθεύουμε τη 16. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 17 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 18 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 19 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 20 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 21 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 23 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 25 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 26 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Και φτάνουμε στις τρεις τελικές προφορίες. Τελική ψηφοφορία για τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν λοιπόν. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίθηκαν. Το νομοθετικό ψήφισμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία. Πέρας. Ε, αρχίζει, συγγνώμη. Τελική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία και πέρας. Αν ψήφισε και τελευταίος, εγκρίθηκε λοιπόν και συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Μπούζεκ. okay. okay. We usually this and it becomes red. Uh, dear Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ένα πολύ σημαντικό σημείο να εξετάσουμε η συγκίτρια η μία πέτρα να ξέρω ότι είστε αστέρι αγαπητοί συναδελφοί, παρακαλώ κάντε ησυχία για να ξεκινήσουμε αυτή τη σημαντική συνάντηση, πολύ σημαντική, το η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Νεολαίας Συμμετέχονται στο, European Youth Event είναι εδώ. Ο Μπάρι Νουβίνα εδώ κοντά μου. Ο Βενέρεντα δίπλα του. Και ο κύριος Αντρέα Λετσίκονα. τον έχει κύριε Αντρέα -hmm. Α, ο Αντρέα, α, μάλιστα. ο Ανδρέα Ντετσίκο Ναρντόνε. Μπορείτε να μου βοηθήσετε. Ανδρέα Ντετσίκο Ναρντόνε είναι το όνομά μου. Οι ιδέε λοιπόν φέρνουν αυτοί οι νέοι άνθρωποι που μπορεί να είναι ενδιαφέρουσε για το, δικό μα έργο για την, για την έρευνα, την καινοτομία, την ε, ψηφιακή ενιαία αγορά, την ενέργεια, ε, είναι μια σημαντική, σημαντική εκδήλωση που έγινε 20 με 21 Μαΐου 2016 στο Στρασβούργο του χρόνου και πάλι στο Στρασβούργο βέβαια θα γίνει η ίδια εκδήλωση 7.500 νέοι άνθρωποι συζήτησαν όλες αυτές τις ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης η συνάδελφος, η κυρία Σάντερ και ο κύριος Μαντέρ που είναι και ο κύριος Μαρτά μάλλον ο κύριος Μαρτά είναι εδώ δηλαδή η κυρία Σάντερ δεν τη βλέπω πάντως δύο εξ αυτών συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για την Νεολαία να πω δύο λόγια για τους νέους αυτούς ανθρώπους που είναι μαζί μας σήμερα. Ο κύριος Μπάρι Οβίνο Γεννήθηκε το 1991 στο Ναϊρόμπι, στην Κένια. Τον 20ο αιώνα, έπασε, όχι τον 21ο, έτσι. και ήταν εξαιρετικά δραστήριος στην Ευρώπη. Έλαβε πολλά βραβεία δημιούργησε δύο, οργαν... δύο επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων και το Business Breakfast και πολλά άλλα project, project ασχολήθηκε με ζητήματα διεθνούς ε, φορολόγησης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, και εξειδικεύτηκε περαιτέρω στον τομέα αυτών, πολύ κοντά στις δικές μας δραστηριότητες. Η Χέλεν Νερά, 19 ετών, έτσι, όταν κάποιος είναι κάτω από 20, μπορεί να λέμε πια την ηλικία νομίζω, σπούδασε οικονομικά στη Βιέννη, συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων, στην Επιτροπή Ήτρε, καθώς ήταν επίσης και πρέσβης εκπαίδευσης, έχει εμπειρία σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, σε διάφορες επιχειρήσεις, και στην Αυστρία και αλλού. Δραστηριοποιείται λοιπόν στην Ευρώπη σε πολλούς τομεί Και τώρα ο Ανδρέα Λετσίκο Ναρντόνιο που γεννήθηκε στη Ρώμη το 1985 είναι φοιτητή ε, μηχανικός και είναι συμμετέχει σε προβλήματα εκλεκτικής μάθησης είναι υπέρ μιας ε, οριζόντιας ε, διατομιακής προσέγγισης στην εκπαίδευση. Είχε πάντα πάθος με την οικονομία και την πολιτική πώς αυτά, αυτοί οι δύο τομείς μπορούν να βελτιώσουν το βιωτικό επίπεδο της κοινωνίας και θέλει να γίνει επιχειρηματίας ε, για να βοηθήσει θα να αναπτυχθεί περαιτέρω η Ευρώπη. Αυτά λέει και το βιογραφικό σα νομίζω. Λοιπόν, προτείνω σε μια πρώτη φάση για την έρευνα και την καινοτομία ορίζοντα 2020. Θα μιλήσουμε, θα δώσω το λόγο σε δύο από εσά. την Ελένα και τον Αντρέα. Δύο λεπτά ο καθένας να μας παρουσιάσετε μία ιδέα. Πρώτα η Έλενα και μετά ο Ανδρέα. Και μετά μπορώ να δώσω το λόγο σε κάποια μέλη αν θέλουν να ρωτήσουν οτιδήποτε ή αν έχουν σχόλια. Και θα έχετε μετά ένα, λεπτό για να απαντήσετε, να αντιδράσετε. Αυτά για την πρώτη ενότητα. Στη δεύτερη ενότητα θα μιλήσουμε για την κυβερνοασφάλεια και την ενιαία ψηφιακή αγορά και μετά θα μιλήσουμε και για την ενεργειακή ασφάλεια μια τρίτη ενότητα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ελένα και Ανδρέα. Αλλά και ο Μπέρι στη συνέχεια όμως. Ελένα, δύο λεπτά. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ιδέα την οποία θέλω να σας παρουσιάσω είναι να κάνει μια να είναι πιο ελκυστική η καριέρα στον τομέα της έρευνας για ε, τουλάχιστον πέντε έτη μετά την αποφύτιση. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται ένας δρόμος της αδειοδρομίας με συγκεκριμένε προοπτικές για νέους επαγγελματίε για πέντε χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ε, πρόγραμμα έρευνας στα πλαίσια του 2020. Αυτές οι μελέτες έρευνας θα, θα πρέπει να γίνει μια έρευνα για να δούμε πώς οι βιομηχανίες και τα ερευνητικά κέντρα συνεργάζονται για να ε, καταλάβουν καλύτερα την παρούσα κατάσταση. Από εκεί πέρα θα πρέπει να δημιουργηθεί μια προδιαγραφή για να μπορούν οι νέοι άνθρωποι να περάσουν από τις επιχειρήσεις ε, στις, ε, στις, στο πανεπιστήμιο. Συνήθως η χρηματοδότηση είναι στην, στην πρώτη γραμμή. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να μπορούμε να αναπτύξουμε όμως και τους ανθρώπινους πόρους για να μπορεί να λάβει χώρα η έρευνα και αυτή η διαδρομή που θέλω να προτείνω εγώ ε, θα μπορούσε στην αρχή της καριέρας ενός ερευνητή ε, να υπάρχει εναλλαγή από το πανεπιστήμιο προς την επιχείρηση. Αυτή η εναλλαγή θα μπορούσε να γίνει και σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Ε, θα, μπορούσαν, θα μπορούσαν να έχουν, να έχουν παρεμφερούς, παρεμφερείς μισθούς και κοινωνικές, κοινωνικά επιδόματα. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις συνθήκες εργασίας, την παραγωγικότητα, να δοθούν κίνητρα ε, στους διάφορους ακαδημαϊκούς οργανισμούς ε, και να τους συγκρίνουμε με το τι συμβαίνει σε ιδιωτικό επίπεδο, σε ιδιωτικών επιχειρήσεων. Θα πρέπει να δούμε ε, πώς λειτουργεί αυτή η πρακτική των βραχυπρόθεσμων συμβολέων έρευνας και το πώς αυτό και κατά πόσο τελικά αυτό είναι υποφέρει για τι επιχειρήσει. Πρέπει να έχουν αφροπτικοί προοπτική ερευνητέ στην αρχή τη καριέρα του για λόγου κοινωνική ασφάλεια, διότι δεν θα έχουμε, έχουμε πολλού τέτοιου στο μέλλον. Ελπίζω αυτή η πρόταση να είναι χρήσιμη. Ευχαριστώ. Εγώ πίστευα ότι θα μιλήσετε 3-4 λεπτά, αλλά πραγματικά σεβαστήκατε το χρόνο. Θέλαμε να δούμε ε, τι μπορεί να πει κανεί τελικά σε δύο λεπτά, παρουσιάζοντα μια νέα ιδέα. Πολύ ωραία. Ο Ανδρέα τώρα. Παρακαλώ, μια πρόταση με την ιδέα σου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, αναγνωρίζω ότι στο σύστημά μας ε, εκπαιδεύουμε αυτή τη στιγμή το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος. Ξέρουμε ότι οι κοινωνίες αλλάζουν γρήγορα. Οι νέοι λοιπόν πρέπει να έχουν ε, καινούργια προσόντα, καινούργιες δεξιότητες, τα οποία δεν είναι ακόμα ενσωματωμένα στα συστήματα εκπαίδευσης. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να φέρουν ε, αυτά τα, αυτές τις δεξιότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα. Πρέπει να γίνει μια μελέτη λοιπόν για το πώς οι εταιρείε και οι βιομηχανίες ε, διαδρούν με ε, το εκπαιδευτικό σύστημα και πώς, πώς μαθαίνουν στα σχολεία τα των επιχειρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν να εξεταστούν διτές προσεγγίσεις. Θέλουμε να δημιουργήσουμε λοιπόν με τη μελέτη αυτή αφενό ένα κοινό τρόπο ώστε οι επιχειρήσει να έρθουν σε διάδοση με τη σχολεία, ε, με εργαστήρια, ε, με ε, συγκεκριμένα μαθήματα και να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση που να δίνει στου Ευρωπαίου μαθητέ τι ίδιε ευκαιρίε. Για να έχουν τι ίδιε ευκαιρίε πρέπει να έχουν και την ίδια προετοιμασία, την ίδια κατάρτιση. Χρειάζεται λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν κάποιες κοινέ δεξιότητες στην Ευρώπη. Χρειάζεται αυτή η συνεργασία μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων. Ανά την Ευρώπη οι νέοι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες, τις ίδιες πιθανότητες. Και θα πρέπει το σχολείο να έρθει κοντά στις επιχειρήσεις, αλλά και οι επιχειρήσεις να έρθουν κοντά στο σχολείο. Είναι ο μόνος τρόπος για να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία, ε, τα αυτά που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις, και κατάλληλες γνώσεις ε, που απαιτούν ε, οι εταιρείε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εκπληκτικό το αποτέλεσμα. Εμείς μέρες φορές ε, κάνουμε μιλήσει ενός λεπτού που δεν αρκεί, αλλά για εσάς τα δύο λεπτά είναι πολλά από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, ευχαριστώ για την εισαγωγή σας για την παρουσίαση της ιδέας σας. Το πρώτο αφορούσε τη βελτίωση των στα σταδιοδρομίας για τους νέους, ιδιαίτερα τις γυναίκες. Δεν νομίζετε ότι ισχύει γι' αυτό. Και το θέμα της ε, ενσωμάτωσης ε, της εκπαίδευσης με τις μελλοντικές ε, ε, προοπτικές στην αγορά εργασία. Λοιπόν, ε, ο κύριος Μαρτάν που ήταν στη συνάντηση στο Στρασβούργο, θέλετε να πείτε δύο λόγια. Εσείς δεν έχετε όριο χρονικό. Όχι, δεν υπάρχει όριο. Ευχαριστώ Πρόεδρε κάθε φορά που μου δίνετε το λόγο μου λέτε ότι πρέπει να σέβομαι το χρόνο. Ε, θα προσπαθήσω. Ήθελα να υπογραμμίσω ότι ναι, όντως για τρίτη φορά συμμετείχα σε αυτή την εκδήλωση που είναι πραγματικά καταπληκτική. Έχουμε πολλά να μάθουμε από τους νέους. Πρέπει να απαντάμε στα ερωτήματα που θέτουν και πραγματικά ε, με πικρία βλέπω ότι μας θέθηκαν μια σειρά από ερωτήματα από όλους τους νέους που ήταν εκεί εμείς αυτές τις ερωτήσεις τις διαβάσαμε στην Επιτροπή και ακόμα δεν έχουμε απαντήσεις. Ε, ένα ελάχιστο λοιπόν δείγμα σεβασμού είναι να απαντάει κάποιες ερωτήματα που του θέτουν στην Δημοκρατία. Τώρα, το να γίνει η σταδιοδρομία, η επιστημονική, η ερευνητική, πιο συναρπαστική. Συμφωνώ απόλυτο. Είχα πάει σε μέρε πολιτείε πριν από μερικά χρόνια και είδα ότι εκεί υπάρχουν πολλά μέσα διατίθεται πολλά μέσα έτσι ώστε οι σταδιοδρομίε στον τομέα της έρευνας, ε, στον τομέα των επιστημών να είναι συναρπαστικές. Πολλοί λοιπόν έρευνητές πάνε εκεί διότι εκεί τους δίνουν τα μέσα ε, για να κάνουν τη δουλειά τους. Βεβαίως ε, υπάρχουν κάποια πράγματα στην Ευρώπη, υπάρχουν οι δράσεις Marie Curie, υπάρχουν υποτροφίες για την έρευνα, μπορεί κάποιος να χρηματοδοτήσει ένα διδακτορικό σε μια επιχείρηση, αλλά πρέπει να υπογραμμίσω ότι το θέμα είναι πώς θα αυξηθούν τα μέσα, ο κοινωνικός προπολογισμό για να μπορούν οι νέοι άνθρωποι αυτοί να μένουν στην Ευρώπη και να κάνουν εκεί την καριέρα τους. Θα πρέπει από την άλλη να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο και τις επιχειρήσεις που ορισμένε φορές περιμένουν πολλά από τη, τα δημόσια κονδύλια. Κάτι που δεν συμβαίνει στις ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούν τα πανεπιστήμια θεωρώντας ότι αυτό είναι μια επένδυση. Αναμένουν να την αποσβέσουν κάποια στιγμή. Ενώ στην Ευρώπη οι επιχειρήσεις θέλουν άλλοι να επενδύσουν για αυτούς. Και αναμένουν όμως αυτοί οι ίδιοι να αποκομίσουν τα ωφέλη. Με ενδιαφέρον λοιπόν να πω ότι συμμερίζομαι, ε, συμμεριζόμαστε ουσιαστικά τα ίδια ε, ψήφισε ανησυχίε για το πώ θα μείνουν οι Ευρωπαίοι ερευνητέ στην Ευρώπη και πώ θα δημιουργηθούν πραγματικέ συμπράξει να ε, περάσει και στην οτροπία των ενδιαφερομένων ότι μπορεί κανείς εύκολα να περνάει από τι επιχειρήσει ε, ε, στα πανεπιστήμια και στην εκπαίδευση και τούμπαλιν. Σα ευχαριστώ για τι τις σα. Μάλιστα. Και τώρα ο Ρόιλ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, σύντομες αλλά γεμάτες ενδιαφέρον και περιεχόμενο αυτές τις παρεμβάσεις. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω την εξή ερώτηση. Βλέπουμε πολύ συχνά οι νέοι να μας λένε, αντίθετα από ό,τι πολλούς φορέ από πεπειραμένους πολιτικούς, ότι πρέπει να συνδυαστεί η εκπαίδευση με την επαγγελματική κατάρτιση, με την προετοιμασία για τον επαγγελματικό βίο και ότι δεν έχει κανένα νόημα να κάνει κανείς σπουδές οι οποίες όμως δεν είναι χρήσιμες για την επαγγελματική ε, ανέληξη στη συνέχεια. Τα κράτη τα οποία έχουν κάνει την επιλογή αυτή του διοδικού συστήματος έχουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας μάλιστα. Αυτό βλέπουμε ότι να το αγνωρίσουν οι νέοι. Πώς μπορούμε πιο συγκεκριμένα να το κάνουμε ε, έτσι ώστε να καταλήγει αυτή η διαδικασία της εκπαίδευσης σε μια θέση εργασίας και εσείς πώς συγκεκριμένα το αξιολογείτε. Και δεύτερη ερώτηση Πολύ συζητούμε για την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, τους κινδύνους που μπορεί να συνεπιφέρουν. Εσείς αντίθετα όμως μας λέτε ότι μπορούν να αποτελέσουν μια μεγάλη και σημαντική ευκαιρία. Αυτά δηλαδή τα οποία ε, θα μας φέρουν στο μέλλον πρέπει να στηρίζονται πάνω στην εφαρμογή της καινοτομίας και της τεχνολογίας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το μέλλον. Πολλές φορές όμως το φρένο το τραβάει η πολιτική και δεν επιτρέπει στην, ε, σε ένα νέο σχέδιο καινοτόμο τεχνολογικά να υλοποιηθεί. Θα θέλατε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Τσόκα έχει τώρα τον λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους νέους ε, για αυτές τους, ε, τις προσπάθειες και ιδιαίτερα και για την έμφαση στο θέμα αυτό που είναι πολύ σημαντικό, την ανάλυση στην οποία προβαίνεται, που είναι πολύ σημαντική σχέσεις πανεπιστημίου επιχειρήσεων, έρευνα ε, βασική και εφαρμοσμένη, έρευνα και παραγωγή. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω μετά τη διάγνωση και τις τοποθετήσεις σας, που βέβαια τείνουν και προς το αίτημα της ενίσχυσης των πόρων για την έρευνα, θέλω να ρωτήσω τι είδου ε, μοχλό υποστήριξης, μόχλευσης θα μπορούσαμε να δούμε στην ε, αποφορολόγηση, στην μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης ε, στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να επενδύουν στους τομείς αυτούς, χάρη στον περιορισμό της ε, φορολογίας. Ευχαριστώ. Κύριο Ευχαριστώ τους ε, νέους μας. Ιδιαίτερα με ενδιαφέρον άκουσα την ε, τοποθέτηση για την εκπαίδευση από τον ε, συμπολίτη μου. Θέλω βέβαια να πω ότι υπάρχουν πολιτικές και κυρίως η πολιτική της λιτότητας οι οποίες καταστρέφουν τη δημόσια εκπαίδευση σε πολλές χώρες και σε όσο συμφωνώ ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού, της επιχείρησης, του ιδιωτικού τομέα της επιχείρησης, της δημόσιας εκπαίδευσης δεν θα πρέπει αυτό να υποκαταστήσει τη δημόσια και κρατική εκπαίδευση και η οποία θα μας επιτρέπει να εργαζόμαστε σε όρους ελευθερίας. Γιατί ενσυχώ ιδιαίτερα για την κατάσταση των σχολείων στην Ιταλία όπως και στην Ελλάδα. Ξέρω ότι οι διεθνείς ανταγωνιστές, η Κίνα παραδείγματι, έχουν εγκρίνει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για τον τομέα της εκπαίδευσης, ενώ εμείς δεν έχουμε ούτε καν wifi και ίντερνετ στα σχολεία μας. Θα πρέπει λοιπόν Εάν θέλουμε η Ευρώπη να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της, να αρχίσουμε να επενδύουμε με σοβαρότητα στους νέους και να μην κάνουμε ζημιά στην ίδια την εκπαίδευση με τις πολιτικές αυτές που φέρνουν καταστροφικά αποτελέσματα. Κόχλετσεκ. Protože jsem si bral řadu eh, studenty z jako diplomanty. Πρόεδρε, Και εγώ έπαιρνα ε, ε, εκπαιδευόμενο, μαθητευόμενο στην εταιρεία που εργαζόμουν πριν από χρόνια και συχνά εντυπωσιάστηκα από το ενδιαφέρον του και από αυτά που ήθελαν πραγματικά να μάθουν. Αυτό που ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον ήταν το ότι αναρωτιόνταν αν η, εκπαίδευση μέχρι το, το πτυχίο, μέχρι μάλλον ε, το ε, πρώτο πτυχίο, ε, αρκεί και αν θα έπρεπε να έχει μια πρακτική απασχόληση, μια εξάσκηση και ακόμα και αν κάποιος θέλει να γίνει ερευνητής να έκανε πρώτα κάτι το πρακτικό. Βέβαια, αν είναι κάτι το θεωρητικό, πάλι μπορεί να έχει και πρακτική εφαρμογή. Και έπειτα, ποια είναι πιο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε να εισαχθεί στα λύκεια. Η ρομποτική, νανοτεχνολογίες, νέα είδη μέτρησης, ε, τι είδου θέματα πιστεύετε, οι σπουδές, η ύλη πιστεύετε ότι θα πρέπει να αρχίσει να διδάσκεται στα λύκεια, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μας λείπουν μόνο η αλλά και οι απόφοιτοι ηλικίου που να ε, είναι αρκετά εκπαιδευμένοι. Κυρία Τόγια. Ευχαριστώ. όπω έλεγε ο συνάδελφο, είναι πολύ σημαντικό αυτό το ραντεβού που ε, παραλαμβάνετε κάθε χρόνο μαζί σας. Πάντα ακούμε πολύ ενδιαφέρουσε ιδέες. Με εντυπωσίασε η ομιλία για την εκπαίδευση και την απόκτηση δεξιοτήτων πιο κατάλληλων για τον επαγγελματικό βίο και ιδιαίτερα το ότι υπογραμμίσατε το σύνδεσμο μεταξύ, την ενίσχυση του ανδεσμού μεταξύ του σχολείου και του επαγγελματικού κόσμου, του πανεπιστημίου και της έρευνας, της βιομηχανίας που εφαρμόζει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας και δίνει τη δυνατότητα για μια τεχνολογική μεταφορά, υλοποίηση που μπορεί να λάβει και βιομηχανικό χαρακτήρα, εν πάση περιπτώσει εφαρμογή τη ε, ε, τεχνολογίες προς το συμφέρον όλων των πολιτών. Είναι ενδιαφέροντα αυτά τα θέματα. Η Ευρώπη σε πολλά κράτη-μέλη υποστηρίζει με κίνητρα που δίνει προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, ιδιαίτερα για την Ιταλία μπορώ να σας πω ότι προσπαθεί με χάρη ε, η Ευρώπη με τις προσπάθειές της να πιέσει προς την σύνδεση του σχολείου με, το με τον επαγγελματικό βίο. Το ίδιο προσπαθούμε και εμείς από εδώ ώστε να ενισχύσουμε τους πόρους ε, για την έρευνα, για την εκπαίδευση και όχι μόνο για τους πρόσφυγες εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι ιδιαίτερα κάνουμε τις προσπάθειες αυτές μέσα στα ε, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πολλές ερωτήσεις ε, επιτάπητος και θα ήθελα να πω στους νεαρούς μας φίλους ότι Έχουμε ε, ακούσει ερωτήσεις από όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί οι συνάδελφοι προέρχονται από διάφορες ε, ομάδες και δεν σας δίνω όριο για τις απαντήσεις, γιατί πήρατε τόσες πολλές ερωτήσεις που θα ήταν άδικο να σας περιορίσω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Με χαρά άκουσα όλα τα ερωτήματα και όλες τα σχόλια για τις δικές μας προτάσεις, γιατί αυτό με κάνει να πιστεύω πως εκτιμάτε τις απόψεις μας και ότι, ε, ότι εισακούγονται αυτές. Τώρα για τις ερωτήσεις. Μία αφορούσε τις καλύτερες σπουδέ. κατά πόσο τα, οι σπουδέ για πρώτο πτυχίο ήταν αρκετά καλέ για την οικονομία και την δίκηση επιχειρήσεων ω ε, φοιτήτρια στην Βιέννη. Είναι αυτό που ε, έχω ω εμπειρία. Βρίσκω ότι οι σπουδές είναι πιο προσιτές για πολλούς και επειδή έχουμε δύο και τρία χρόνια ανάλογα με το πτυχίο και το μάστερ στο Πανεπιστήμιο μου να σας πω ότι είμαστε 23.000 φοιτητές και είμαστε μικρό πανεπιστήμιο της Βιέννης. Η χώρα μας έτσι κι αλλιώς έχει 8 εκατομμύρια κατοίκους. Νομίζω πως αυτό λέει πολλά για την ε, παιδεία μας και για το ε, κατά πόσο αυτή είναι διαθέσιμη για το ανθρώπους από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε ε, όσον αφορά τη θεωρητική έρευνα. Πιστεύω πως οι φοιτητές που μόλις έχουν κάνει ένα διδακτορικό ή ένα μάστερ και που κάνουν έρευνα, δεν είμαι βεβαία κατά πόσο αν τους πείτε να κάνουν εφαρμοσμένη έρευνα ή πρακτική άσκηση θα βελτίωνε τα αποτελέσματα της έρευνάς τους όταν θα επανέρχονταν σε αυτήν. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι στις εταιρείες έχουμε περισσότερη εφαρμοσμένη έρευνα παρά θεωρητική. Και πολύ συχνά οι απόφετοι αποφασίζουν να μην μείνουν στα πανεπιστήμια ή στα ε, ερευνητικά ιδρύματα, αλλά πηγαίνουν στις εταιρείε όπου κάνουν πρακτική έρευνα, φαντάζομαι, που ε, θα λέγεται αυτή. Ωστόσο, ορισμένοι αναγκάζονται να το κάνουν αυτό γιατί δεν υπάρχουν πολλέ εναλλακτικέ, διότι με τα πανεπιστήμια συχνά η μισθή και η κοινωνική πρόνοια δεν συγκρίνονται με αυτά που είναι ο ιδιωτικό τομέα. Επίσης, οι περισσότεροι φοιτητέ που γνωρίζω δεν επιλέγουν την ε, έρευνα γιατί ξέρουν πόσο δύσκολο είναι το, η διαχείριση της έρευνας. Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει κανείς να αγωνιστεί για να μπορέσει να κάνει την έρευνά του, ενώ στον ιδιωτικό τομέα είναι πιο εύκολο ε, και γι' αυτό δεν έχουν εναλλακτική περισσότερη εφαρμοσμένη έρευνα, βέβαια, προέρχεται από τη θεωρητική. Ε, περισσότεροι που εγώ τουλάχιστον γνωρίζω είναι ότι θέλουν να κάνουν εφαρμοσμένη έρευνα και η θεωρητική έρευνα αφήνεται στους ανθρώπους που συμφωνούν και δέχονται να αγωνίζονται καθημερινά για να στηρίξουν την έρευνα τη θεωρητική τους, δέχονται τους μισθούς και τις, ε, την κοινωνική πρόνοια που τους δίνεται και δεν ξέρουν καν αν του χρόνου θα μπορούν να συνεχίσουν την έρευνα αυτή. τελευταία ερώτηση, ποιο είναι το πιο σημαντικό θέμα. Το πιο σημαντικό θέμα που πρέπει να μπει στο Λύκειο, η διδακτέα ύλη, είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση γιατί πρόσφατα έμαθα από τους συναδέλφους ότι στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει θέμα critical thinking, κριτική σκέψη. Δεν το είχα ξανακούσει ποτέ αυτό πριν, αλλά νομίζω πως είναι ένα από αυτά τα θέματα όπου δεν μαθαίνεις γνώση απαραίτητος, αλλά δεξιότητες ώστε να μπορείς μετά να αποκτήσεις γνώση ο ίδιος. Είναι πολύτιμο αυτό, γιατί όταν, ε, γιατί όταν τελειώσει το σχολείο και το πανεπιστήμιο, δεν θα έχεις κανέναν δάσκαλο μπροστά σου ή καθηγητή να σου λέει τι πρέπει να μάθεις, θα πρέπει να μάθεις μόνος σου και θα χρειαστεί να έχεις τις απαραίτητες δεξιότητες για να το κάνεις αυτό. Οι δεξιότητες λοιπόν όπως η κριτική σκέψη είναι πάρα πολύ σημαντική και εγώ θα ήθελα τα δικά μου παιδιά να μάθουν τέτοια πράγματα στο σχολείο. First να πω στην κυρία Τόγια ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να γίνονται επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά όπως είπατε, δεν μιλάμε για το τι κάνουν τα κράτη-μέλη, θα έπρεπε να μιλήσουμε για το τι κάνει η Ευρώπη, γιατί δεν είμαστε μόνο μια κοινότητα. Ε, συχνά όταν μιλάμε για τους νέους, να ξέρετε ότι εμεί αισθανόμαστε Ευρωπαίοι, δεν πρέπει να μοιραζόμαστε μόνο τις αξίες, αλλά και την προετοιμασία και τις δυνατότητες. Γι' αυτό έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μοιραζόμαστε. Δεν είμαστε από την Ιταλία, δεν είμαστε από τη Γαλλία, δεν είμαστε από τη Γερμανία. Αυτό είναι ο τρόπος να προχωρήσουμε και να ε, προωθήσουμε αυτή την αίσθηση κοινότητας. Το τι θα πρέπει να διδάσκεται τώρα στα σχολεία, όπως ρώτησε ο κ. Κόχλιτσεκ, ιδιαίτερα στα Λύκια. Εμένα η δική μου ιδέα, το να έχουμε μια μελέτη για το τι γίνεται, μάλλον το τι γίνεται, η σύνδεση ανάμεσα στη βιομηχανία και την ε, παιδεία ε, πρέπει να ξεκινά από τα λύκεια, γιατί ακριβώς τα λύκεια πρέπει να διδαχθούν οι ε, δεξιότητες που ο κόσμος θα χρειαστεί για το μέλλον, που τα παιδιά θα χρειαστούν για το μέλλον, θα χρησιμοποιήσουν στην πράξη για το μέλλον. Και πρέπει αυτό να το μαθαίνουν, να μην μαθαίνουν μόνο θεωρίες και καλύτερες πρακτικές, αλλά και κοινωνικές πρακτικές, γιατί στον αυριανό κόσμο θα χρειαστεί να έχεις ε, ικανότητες για προγραμματισμό, οι υποστημονικές δεξιότητες, γιατί στο μέλλον όπως είπε και ο κύριος Ρόιλ, να, να, να μην μας φοβίζει το μέλλον. Δηλαδή, το εργατικό δυναμικό δεν θα ασχολείται μόνο με μηχανήματα ή να κάνει επαναληπτικές εργασίες. Ακόμα ίσως και ένας δημοσιογράφος να μην είναι δουλειά του μέλλοντος, χάρη στην τεχνητή ευφυΐα. Αλλά αυτό δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Πρέπει να προχωρήσουμε με αυτό, να το επιτρέψουμε και να το ε, να το δεχτούμε. Γιατί όταν αυτό θα συμβεί θα μείνουμε εμείς πίσω. Εμείς χρειάζεται να δράσουμε τώρα, όπως έκανε η Apple, ας πούμε, που απέρριψε τελείως το, το, το τελευταίο iPhone, γιατί είναι αυτοί που έχουν τη νέα τεχνολογία και θα είναι οι πρώτοι που θα φτιάξουν κάτι νέο. Τώρα πρέπει να επενδύσουμε στους νέους γιατί στο μέλλον δεν θα είναι εργάτες, θα είναι δημιουργοί, θα είναι προγραμματιστές, θα είναι άνθρωποι που θα φτιάχνουν πράγματα. Δεν θα είναι αυτοί που θα συναρμολογούν απλά πράγματα. Και αυτό πρέπει να το προβλέψουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μέσο όρο ανθρώπων ε, χωρίς δεξιότητες. Πρέπει να τους μάθουμε να μπορούν να δημιουργήσουν, γιατί διαφορετικά όλα ε, η εξυπνάδα, η ευφυία ευρωπαϊκή, ο πολιτισμός ευρωπαϊκός θα μείνει πίσω. Γιατί θα έρθουν οι Κινέζοι που έχουν τους εκτυπωτές τους τρισδιάστατους, ξέρουν να τους χρησιμοποιούν και ξέρουν να φτιάχνουν πράγματα. Και θα έχουν αυτές τις ικανότητες, τις δεξιότητες που εμείς έχουμε μείνει πίσω. Δεν πρέπει να μένουμε στην, και να κολλάμε στην παλιά νοοτροπία πριν από 20 χρόνια, γιατί ο κόσμος αλλάζει κυρίως με τα κοινωνικά μέσα και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το διδάσκουμε, να διδάσκεται. Γιατί όταν μιλάμε για ασφάλεια στοιχείων, δεδομένων, που είναι πάρα πολύ σημαντικά οι νέοι, κυρίως οι νέοι, δεν έχουν ιδέα. Και γίνει και αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο καθημερινά. Γιατί δεν ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Πρέπει λοιπόν ένα μάθημα να τους μαθαίνει πώς θα έρχονται σε επαφή με αυτό το νέο κόσμο. Όχι με τις δεξιότητες πριν από 10 χρόνια, που ήταν τελείως διαφορετικός ο κόσμος. Και όταν μιλάμε για που ρώτησε ο κύριος Τσόγκα για την ε, φορολόγηση των εταιριών. Η φορολόγηση χρησιμοποιείται και για την παιδεία η παιδεία θα έπρεπε να συνεργάζεται με τη βιομηχανία, με, με τις επιχειρήσεις. Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν και να επενδύσουν στην έρευνα. Να δημιουργείται έτσι ένα έφορο περιβάλλον για τι επιχειρήσει. Σω α πούμε να δίνεται κάποια φοροαπολογία όταν επενδύουν οι επιχειρήσει στην έρευνα, στα σχολεία και, στις, ε, και στα πανεπιστήμια, ώστε να μπορούν εκείνοι να προχωρούν περισσότερο. Δηλαδή να υπάρχει συνεργασία, συνεννόηση, συντονισμός. Χρειαζόμαστε δηλαδή παρακολούθηση από τη μια πλευρά τη φορολόγηση και από την άλλη πλευρά ε, να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, νεαροί μου φίλοι. Ε, Για αυτή τη συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και τώρα πάμε στη ψηφιακή ενιαία αγορά. Μπάρι, δύο λεπτά. Και μετά θα ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Η πρώτη μου ιδέα είναι να εγγυηθούμε αδιάκοπτη διασύνδεση στο ίντερνετ σε όλες τις ευρωπαϊκές ε, πόλεις, καθώς και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων, γιατί εκεί συναντώνται κάθε είδους άνθρωποι για, να, ε, για επαφές, για εμπόριο ή οτιδήποτε. Η κινητικότητα είναι πυλώνα τη Ευρωπαϊκή Δομή, και γι' αυτό πρέπει οι δημόσιοι χώροι να είναι ασφαλισμένοι απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και τις τρομοκρατικές απειλές. Σε δύο τρόποι υπαρχουν ε, υπάρχουν. Δηλαδή, ε, δωρεάν Wi-Fi στις δημόσιους χώρους και τις δημόσιες μεταφορές, γιατί ε, κάτι τέτοιο μπορεί γρήγορα να ελεγχθεί από τις δημόσιες αρχές σε περίπτωση επίγουσας ανάγκης, αλλά θα είναι και δυνατόν να ειδοποιηθούν οι δημόσιες αρχές σε περίπτωση κινδύνου ή κάποιου έκτακτου γεγονότος. Δεύτερον, να υπάρξει κοινή εφαρμογή για όλα τα κρατημέλη που να εγκαθίσταται σε όλα τα εφή τηλέφωνα, οι αστυνομικές αρχές και οι τοπικές αρχές να στέλνουν ειδοποιήσεις συναγερμούς στους χρήστες των smartphone σε δύο γλώσσες, τις γλώσσες, τη γλώσσα της χώρας κάθε φορά και τα αγγλικά, ώστε να δίνονται ε, ε, και οι ε, οδηγίες για τον χρήστη του τηλεφώνου θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για διάφορα θέματα, ας πούμε να ζητηθούν μάρτυρες, ε, ε, αυτόπτες μάρτυρες, εντοπισμός ενός υπόπτου ή ε, κάποιου φυγά. Υπάρχουν εκατομμύρια εφή τηλέφωνα σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα μπορούσαν να επιτρέψουν να συμμετέχουν εκατομμύρια Ευρωπαίοι στην εφαρμογή αυτή, στο app αυτό για την ευρωπαϊκή ασφάλεια θα μπορούσε κάτι τέτοιο να βελτιώσει και για τους, τις δυνατότητες για τους ε, όσους ταξιδεύουν στις διάφορες χώρες και θέλουν να αποφύγουν ε, το ε, υπερβολικό κόστος ή τη χρέωση της περιαγωγής. Θα πρέπει να υπάρχει διαρκής προστασία των πόλεών μας και των πολιτών μας, καθώς και της ποιότητας της ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Chair. Έλενα πάλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δεύτερη μου ιδέα όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και την ψηφιακή αγορά είναι η εξή. Θα ήθελα να υπάρχει νομοθεσία στην Ένωση που ενθαρρύνει τις μη κερδοσκοπικές νεοφυείς ε, εταιρείε τεχνολογίες καθώς και μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή ε, ψηφιακή αγορά. Να μπορούμε να χρησιμοποιούμε το, τις πληροφορίες του ίντερνετ και γνωρίζουμε ότι τα ε, ε, στοιχεία μας θα συλλέγονται και θα πολλούνται. Εμείς φανταζόμαστε κοινωνικούς χώρους όπου μας δίνει την επιλογή να προσφέρουμε τις πληροφορίες μας και όχι να γίνεται αυτό εναγκαστικά επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική. Όταν μας να ε, κλικάρουμε σε ένα κουμπί για να, για να συμφωνήσουμε για το να δοθούν οι πληροφορίες μας. Δεν έχουμε συνήθως επιλογή γιατί ε, δεν υπάρχει άλλο δίκτυο ή είναι ένα άλλο δίκτυο μόνο υπάρχει το οποίο είναι πολύ λιγότερο δημοφιλές. Όταν ε, συμφωνείς λοιπόν να φτιάξεις το δικό σου λογαριασμό, συμφωνείς είτε για να χρησιμοποιεί τα στοιχεία σου είτε διαφορετικά δεν μπορείς να χρησιμοποιείς το δίκτυο όπου ανήκουν οι φίλοι σου και η οικογένειά σου. Ε, θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν κατάλληλη νομοθεσία που βοηθά σε αυτέ τι περιπτώσει και μα επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα ακόμα και αν δεν θέλουμε οι πληροφορίε μα να δίνονται. Ε, να δημοσιεύονται. Επίσης θα ήθελα να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσει σε νομοθεσία με κοινού κανόνες ώστε να μην υπάρχουν 28 διαφορετικές ψηφιακές αγορές και να στηριχθούν οι μη κερδοσκοπικέ εταιρείε. γιατί ο ψηφιακό χώρο δεν θα, θα πρέπει να είναι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει τι νεοφύης εταιρείε λοιπόν αλλά και να έχουμε και ένα είδος καλύτερης δυνατή εταιρεία ώστε να μπορέσει να ε, έχει ανωδική πορεία και η αγορά ε, εργασία, αγορά μας. Θα μπορούσε έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει στις 20 ε, πρώτες εταιρείε τεχνολογίας, ψηφιακής τεχνολογίας, γιατί τώρα δεν υπάρχει ούτε μια ευρωπαϊκή εταιρεία στις 20 μεγαλύτερες εταιρείε του κόσμου. Αυτά, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Και τώρα παρακαλώ τους συναδέλφους να λάβουν το λόγο, εάν έχουν κάποια ερώτηση. Κύριος Μαχτά, παρακαλώ. Μερικές παρατηρήσεις μόνο. Βέβαια στον κόσμο του διαδικτύου, της σύνδεσης των πάντων με τα πάντα, συμφωνώ μαζί σας ότι η δημιουργία hotspots ή πάντως δημόσιων χώρων με δωρεάν wifi είναι μια ιδέα η οποία προωθείται σε πολλές χώρες. Στην πατρίδα μου τη Γαλλία υπάρχουν στις ε, μεγάλες πόλεις ζώνες με δωρεάν ε, ασύρματο διαδίκτυο. Βέβαια οι εφαρμογές ασφαλείας είναι επίσης μια πολύ καλή ιδέα, δεδομένου ιδιαίτερα του, δεδομένων των συνθήκων και ιδιαίτερα δεν θέλω να σταθώ στις διακρίσεις εκεί δηλαδή που δεν είναι επαρκώς παρούσα η Ευρώπη ή τα κράτη, περιοχές ολόκληρες όπου δεν υπάρχει καν ίντερνετ υψηλή ταχύτητα, για να μην μιλάμε για, ίντερνετ, για Wi-Fi. Νομίζω ότι υπάρχουν περιοχές που δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει Wi-Fi και εκεί πρέπει η Ευρώπη να επενδύσει ώστε και τα 500 εκατομμύρια των πολιτών της Ευρώπης να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία. Κάτι άλλο που βέβαια δεν θα σταθώ ιδιαίτερα, είναι ότι δεν έχουν όλοι ευφυέ τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό υπολογιστή στη θέση του. Α μην συγχαίουμε λοιπόν το δικαίωμα, την πρόσβαση μάλλον στην πληροφορία και το δικαίωμα στη γνώση και να πιστεύουμε ότι περνάει μόνο μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί αυτό σημαίνει ότι αφήνουμε στο περιθώριο κομμάτι ολόκληρο των, ε, ολόκληρο των πολιτών μα. Βεβαίω πρέπει να γίνει μια προσαρμογή και σύμφωνα σε αυτό για τις νεοφύης επιχειρήσεις. Συμφωνώ, είναι μια συζήτηση που έχουμε κάνει και στο Στρασβούργο. Πολλοί ήταν οι νέοι που μίλησαν για τη δυσκολία της δημιουργίας μιας νεοφύους επιχείρησης στην Ευρώπη, ιδιαίτερα γραφειοκρατία, φορολογία που ξέρω τις ορισμένες χώρες, όπως η δική μου πατρίδα. Ε, μπορεί με το που ιδρύεται μια επιχείρηση και με μηδενικό κύκλο εργασιών να πέφτουν οι φόροι και να πρέπει να πληρώνει κανείς φόρους Επομένως θα πρέπει να δώσουμε ένα περιθώριο, ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια ε, που θα επιτρέψουν ε, στην πρωτοβουλία της νεοφυούς επιχείρησης να επιβιώσει και να αρχίσει να παράγει κέρδος και μεταφόρο. Ε, για το δημόσιο πεδίο επίσης, και επειδή και λόγω ηλικίας δεν γνωρίζω πολλά πράγματα στον, για τον μη εμπορικό τομέα, άλλωστε προερχόμαι από το χώρο της βιομηχανικής παραγωγής, ε, θα συνεχίσει ασφαλώ ο μη εμπορικό τομέα να αναπτύσσεται και αυτό προς, την, προς τον ε, φίλο Ανδρέα. Ε, εξέλιξη και νέες τεχνολογίες όμως δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν υπάρξει και ισχυρή βιομηχανική βάση. Αν θέλουμε την, τις εφαρμογές πρέπει να υπάρχει και ισχυρή βιομηχανική βάση. Πρέπει και τα δύο να συνδυαστούν. Δεν μπορούμε να μιλούμε μόνο για το ένα ή το άλλο και τα δύο πρέπει να συμπορευθούν. Αν συμφωνείτε βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Θέλω και εγώ να γύρω κάποια ερωτήματα. Αγαπητοί νεαροί φίλοι, έχουμε διερμηνείς από 23 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθισμένους στις καμπίνες. Μπορείτε λοιπόν και για να σας δείξω ότι μπορείτε και εσείς να μιλάτε τη μητρική σας γλώσσα, θα αλλάξω, θα, θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, θα βάλετε τα ακουστικά σας. Και κανονικά ξέρετε ότι μιλάω την αγγλική ίσως, αλλά ακούω τη διερμηνία στη μητρική μου γλώσσα. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε. Λοιπόν, να απευθυνθώ πρώτα στον κύριο κάτι σχετικά με την κυβερνοασφάλεια. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και το θέμα της ασφάλειας. Η ισορροπία μεταξύ των δύο δεν είναι απλό. Διότι είναι κάτι που συνδέεται και με τα ζητήματα γενικότερα άμυνας και ασφάλειας, αυτά που συμβαίνουν στο διαδίκτυο, αυτά που συμβαίνουν με την τεχνολογία του διαστήματος, Μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά για διάφορους σκοπούς. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε μια εποχή όπου το διαδίκτυο ε, μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και οι κακοί, αυτοί που θέλουν να κάνουν κακό στην ανθρωπότητα. Πώς θα το αποφύγουμε λοιπόν αυτό. Πώς θα μπορούσαμε να προστατευτούμε. Θα πρέπει και οι αυτές τις πτυχές να λεφθούν υπόψη. Για την Έλενα έχω ένα άλλο ερώτημα. Αναφέρθηκατε στα κοινωνικά δίκτυα, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Ε, ξέρω ότι υπήρξε ένα ειδικό πάνελ στο Στρασβούργο το Μάιο, το οποίο αφορούσε συγκεκριμένα project. Εσείς παρουσιάσετε δύο συγκεκριμένα project, αν θυμάμαι καλά. Το ερώτημα μου είναι το εξή. Στο διαδίκτυο, τι κάνετε με το λόγο μίσους. Πώς μπορούμε να το αποτρέψουμε αυτό. Διότι εδώ φτάνουμε σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο συζήτηση στη δημόσια σφαίρα. Στα κλασικά μέσα, όπως τα γνωρίζουμε, υπάρχει ένας αυτοπεριορισμός, μια αυτολογοκρισία, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τις ακραίες απόψεις. Στο διαδίκτυο δηλαδή όμω πληροφορούν απόψει τι οποίε δεν υπογράφηκε κάποιο. Ε, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη και δεν μπορούμε να τι ελέγξουμε. Και αυτό δημιουργεί τεράστια ένταση μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ χωρών, εθνών. Ε, οδηγεί λοιπόν σε μια νοσηρή ατμόσφαιρα ε, στο διαδίκτυο. Έχετε ιδέες για το τι θα μπορούσε να γίνει γι' αυτό, διότι ταυτόχρονα δεν θέλουμε να λογοκρίνουμε το διαδίκτυο. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε στην ελευθερία του λόγου, που είναι αξία από μόνη της. Δεν βλέπω να θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις απαντήσεις. Πρώτα, ο Μπέρι. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις και τις ερωτήσεις. Ε, να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα του κυρίου Μαρτά. Θα απαντήσω στα γαλλικά, με και μου τέθηκε στα γαλλικά το ερώτημα σε σχέση με το γεγονό ότι υπάρχουν πολλές πόλεις στην Ευρώπη ε, που έχουν αυτά τα hotspot ε, Wi-Fi ε, και στη Γαλλία και στο Άμστερνταμ. Σήμερα είμαστε στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες δεν υπάρχει τέτοιο hotspot Wi-Fi και αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα ε, για την για του δημόσιου χώρου και την ασφαλεία. Να μην μπορεί κάποιο δηλαδή δωρεάν σε ένα δημόσιο χώρο να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν περιφέρειες στην Ευρώπη που δεν, όπου δεν υπάρχει καν ε, γρήγορο ίντερνετ. Εμείς θέλουμε να επικεντρωθούμε ε, βεβαίως στα σημεία που συναντιόνται οι Ευρωπαίοι. Εγώ ζω εδώ στην Φλάνδρα σε μια φλαμανδική ε, περιοχή ε, όπου δεν υπάρχει ε, συνάντηση μεταξύ Ευρωπαίων, αν θέλετε. Εάν όμως υπάρχει μια κρίση σε μια τουριστική πόλη, αυτό δεν αφορά μόνο τις τοπικές αρχές ή το λόγο κράτος μέρος, αφορά το σύνολο των κρατών μελών. Διότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Γι' αυτό λοιπόν επικεντρωθήκαμε περισσότερο στους μεγάλους δημόσιους χώρους. Σε ό,τι αφορά την ε, σύγκρουση μεταξύ του δικαιώματο στην ιδιωτική ζωή ε, και στα θέματα ασφάλειας και καθώς και ό,τι μπορούμε να κάνουμε με την κακή χρήση του διαδικτύου. Εμείς εδώ επικεντρωνόμαστε κυρίως σε εγκληματικές δραστηριότητες που συμβαίνουν, ε, που συμβαίνουν στην πραγματική ζωή, αν θέλετε, που δεν έχουν σχέση με το κυβερνό έγκλημα δηλαδή. Όταν κάποιος ε, δηλαδή έχει υποπτή συμπεριφορά σε ένα δημόσιο χώρο, ε, να μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει πιο εύκολα και να το διαδώσει αυτό. Δυστυχώς δεν έχω ε, επαρκείς απαντήσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε κατά του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, πώς μπορούμε δηλαδή να προλάβουμε τέτοιες επιθέσεις. Ίσως να πρέπει να Έχουμε καλύτερο εξοπλισμό, περισσότερους ε, αστυνομικούς. Ε, σε πολλά αστυνομικά τμήματα στο Βέλγιο, τη χώρα που ξέρω καλύτερα, είναι πολύ παλιός εξοπλισμός, χρησιμοποιούν παλιές τεχνολογίες, οπότε είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουν ζητήματα εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά την Ευρώπη γενικότερα, φαντάζομαι. Τώρα, ιδιωτική ζωή ε, και ασφάλεια. Είμαστε σε ένα δημόσιο χώρο. Σε ένα δημόσιο χώρο ένας πολίτης ε, είναι λογικό να έρθει σε επαφή με άλλους και να ειδοποιήσει, διότι δεν βρίσκεται στο σπίτι του, στο σαλόνι του. Μάλιστα. Ακούσαμε από το Μπάρι ε, ε, να απαντάει χωρίς ε, περιορισμό χρονικό όπως και οι προηγούμενοι μιλητές πριν, αλλά τώρα θέλω παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Θα αναφερθώ στο ερώτημα του λόγου μίσους και της πρόληψης του λόγου μίσους στον διαδικτύο. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, διότι όπως είπατε δεν θέλουμε αυτός ο χώρος κοινωνικής ανταλλαγής να ε, υπόκειται σε λογοκρισία όπως ε, σημαίνει στις εφημερίδες, διότι τότε ποια θα ήταν διαφορά. Τώρα, τι διαφοροποιεί τα κοινωνικά δίκτυα από τους δημόσιους χώρους έξω στον δρόμο. Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε κάποιος ε, να ξεκινήσει ένα λόγο μίσους ε, στο διαδίκτυο, όταν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό στο δρόμο. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα αυτό, διότι τελικά τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένας χώρος ε, συνάντησης, όπως συμβαίνει και στην πραγματική ζωή. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε διαφορετική μεταχείριση ανθρώπων ε, στο διαδίκτυο από ό,τι στην πραγματική ζωή. Θέλουμε να είναι ασφαλές βέβαια στο διαδίκτυο. Το μόνο το οποίο μπορώ να σκεφτώ είναι εκπαίδευση, η παιδεία ε, σε ό,τι φορά τη συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Το πρώτο βήμα για να έχουμε υπεύθυνου ενήλικες ε, και ενήλικες που να μπορούν να καταλάβουν ποιος είναι ο αντίκτυπος του λόγου μίσους είναι η εκπαίδευση των ανθρώπων αυτών όταν είναι νέοι, όταν είναι παιδιά. Διότι αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν με το διαδίκτυο, με τα κοινωνικά, με τα κοινωνικά μέσα δικτύωση. Είναι λοιπόν σημαντικό να αρχίσουμε νωρί, εάν θέλουμε να είναι υπεύθυνοι ενήλικε αυτοί, ε, θα πρέπει να του το μάθουμε από μικρού. Μάλιστα, σα ευχαριστώ πολύ και για τι απαντήσει σα Τώρα, από τη χρήση της ε, ενέργειας. Ε, Ανδρέα, δύο λεπτά. Θα ήθελα να πω πώς, κατά τη γνώμη μου, μπορούμε να βελτιώσουμε την ευρωπαϊκή προσέγγιση στο ότι αφορά τα έξυπνα ε, δίκτυα. Καταρχήν, οι επενδύσεις δεν πρέπει να αφορούν μόνο κοινά project μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, αλλά για τοπικά project στα διάφορα κράτη-μέλη τα έξυπνα δίκτυα είναι τοπικά συστήματα. Θέλουν να βελτιώσουν τη χρήση της ενέργειας τοπικά. Η επένδυση τοπικό επίπεδο θα αλλάξει την συμπεριφορά του καταναλωτή. Αντί να είναι ε, καταναλωτής απλά ενέργειας, να είναι παραγωγός. Αυτά τα έξυπνα δίκτυα οδηγούν σε χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ε, όπως ε, ηλιακή ενέργεια, η αιωλική ενέργεια. Αυτά τα προγραμματισμένα συστήματα επιτρέπουν και μια ε, πιο ε, έξυπνη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας για να μην έχουμε ε, σπατάλη. Πρέπει βεβαίως να είναι συμβατά μεταξύ τους πρόσφυγα αυτά, πρέπει να πληρούν και κάποια κριτήρια. Αυτή τη στιγμή δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν κανόνες στον τομέα αυτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν κατά τη γνώμη μου πρέπει να θεσπίσει κάποια πρότυπα, ε, κάποια, κάποια μορφή πιστοποίησης έτσι ώστε όλα τα μελλοντικά project να μπορούν να είναι συμφωνά μεταξύ του στην Ευρώπη. Αυτή η εναρμόνιση μεταξύ χωρών και πρακτικών είναι κεφαλαιώδης για να εξασφαλίσουμε το μέλλον αυτού του εγχειρήματο. Διότι είναι ευαίσθητα ζητήματα αυτά. Καλύτερη χρήση των ε, πηγών ενέργεια, για να σεβαστούμε την οζόνη του 2020 και βεβαίω το θέμα τη ασφάλεια των δεδομένων. Ω μηχανικό, θεωρώ ότι σε μερικά χρόνια το πώ βλέπουμε το θέμα της ενέργειας ε, θα είναι διαφορετικό θα είναι διαφορετικό από το μέλλον. Η τεχνολογία μας οδηγεί σε νέες οδούς, τις οποίες δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Ε, θεσπίζοντας λοιπόν πρότυπα και ενθαρρύνοντας επενδύσεις μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτήν την κοινωνική αλλαγή. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Ο Μπάρι, ο Μπάρι είναι ο δεύτερος ομιλητής. Η δεύτερη μου ιδέα είναι να δοθεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε πιλωτικά προγράμματα ώστε να μετατραπούν τα υπάρχοντα κτίρια σε κτίρια τα οποία δεν καταναλώνουν άνθρακα. Πρέπει να σταματήσει η χρήση άνθρακα αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους στόχους για την ενέργεια από το 2020 μέχρι το 2050. Ωστόσο, μεγαλύτερη αντίσταση ε, στην ε, μεταρρύθμιση αυτών των κτηρίων, μετασκευή μάλλον των κτηρίων, προέρχεται από την ε, ε, αντίσταση των ιδιοκτητών. Πρέπει να βελτιωθούν τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, ψήξης θέρμανσης και ούτω καθεξής. Η μετακίνηση λοιπόν σε αυτό το είδος τα κατασκευές θα πρέπει να ξεκινήσει από τα, τα σπίτια χαμηλού εισοδήματος, τις οικογένειες μάλλον χαμηλού εισοδήματος, ώστε να μην υπάρξει φτώχεια και στην ενέργεια. Να βρεθούν λύσεις ώστε να μειωθούν τα αποτυπώματα άνθρακα των κτηρίων και όλα αυτά να είναι προσβάσιμα για όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Τα αποτελέσματα των ε, projects αυτών θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ώστε να σχηματιστεί ένας οδικός χάρτης για τους ιδιοκτήτες και να γίνει ε, να θεσπιστούν ε, ενεργειακά πρότυπα απόδοσης για τις νέες κατασκευές και βελτιωμένα ενεργειακά πιστοποιητικά. Αλλά από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 20,3 δις ευρώ για προγράμματα απόδοσης ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ελλάδα ε, ήταν η πρώτη που έχει ε, εγκρίνει τη σχετική οδηγία γιατί θέλει να προωθήσει την οικονομία της ε, χρησιμοποιώντας και προωθώντας τις πράσινες θέσεις απασχόλησης. Ε, άρα λοιπόν ώστε η ενέργεια που θα παράγεται από τα νέα κτίρια να ε, μπαίνει στο grid, στο, στο δίκτυο και να βρεθούν έτσι λύσεις και για τα νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων. Ευχαριστώ. Έχουμε δύο προτάσεις λοιπόν. και τώρα να ακούσουμε παρατηρήσεις από τους βουλευτές της Ήτρε. Συνάδελφε Μαρτά, ναι, δεν έχω ερώτηση, περισσότερο μια παρατήρηση. Ε, την ανάλυση του και των δύο. Πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες όσον αφορά τις τοπικές επενδύσεις και πιστεύω ότι πρέπει να, και αυτό να το ξεπεράσουμε για να υπάρξουν δυνατότητες ατομικές για τους ιδιώτες να φτιάξουν τη δική τους ενέργεια ε, σύμφωνα και με μια ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά μπάρ, εσείς θέσατε το πρόβλημα. Ποια είναι η προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και αν έχει παραπάνω μέσα και κάνει πολλά για να προσπαθήσει να αναπτύξει την παραγωγή νέου είδους ενέργειας, δηλαδή ανανεώσιμης, υπάρχει πρόβλημα βασικό στο οποίο δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Δηλαδή, πώς θα μπορέσει να έχουν πρόσβαση όλοι χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις σε αυτή τη νέα ε, τα νέα είδη ενέργεια. Υπάρχει το θέμα της ενεργειακής φτώχειας. Εάν είναι αυτό η δυνατότητα στην Ευρώπη, γιατί ας πούμε όταν στα κτίρια χαμηλής κατανάλωση κυρίως είναι, είναι πάντα πιο ακριβά για επενδύσεις και πιο ακριβά να τον νοικιάσει κανείς. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν τα μέσα για τη δημιουργία και την κατασκευή νέων κτηρίων και νέων, νέου είδους θερμικής ε, μόνωσης, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια συνοδευτική κοινωνική πολιτική, ώστε να τα καθιστά προσβάσιμα για προσιτά σε όλους. Ευχαριστώ συνάδελφε. Εγώ έχω μια ερώτηση. Αν μου επιτρέπετε, Smart um, energy electricity. Uh, we discuss very often για την ηλεκτρική ενέργεια. Συχνά μιλάμε για την πρωτοβουλία των Εφιών πόλεων. Θέλουμε επίσης να οργανώσουμε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα τεχνολογίας για τα ΕΦΗ e e δίκτυα. ETP για τα ΕΦΗ e δίκτυα, smart grids. Και ξέρουμε ότι αυτό συμβαδίζει. Δηλαδή η Ενεργειακή Ένωση και η ψηφιακή ένωση. Δεν μπορούμε να έχουμε ασυμμετρικά δίκτυα για τον ηλεκτρισμό χωρίς να αναπτύξουμε και την ψηφιακή μας ένωση, την ψηφιακή τεχνολογία. Είναι αλληλένδετα. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό με αυτή τη τέτοια γενική ε, εικόνα για τις τεχνολογίες και την προώθηση σπιτιών, ε, που δεν καταναλώνουν άνθρακα. Και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Γιατί θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι σε ολόκληρο τον κόσμο η Ευρωπαϊκή Ένωση στην μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ώστε να προστατέψουμε το κλίμα μας. Ακούμε συχνά οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα. Πράγμα που μπορεί κάποιε φορέ όμω να είναι ε, δαπανηρό για τη βιομηχανία μας. Και η βιομηχανία μας να φύγει την Ένωση για να πάει σε άλλε χώρες. Όπου δεν δεν υπάρχουν τόσο ψηλέ προσδοκίε ω προ το κλίμα. Και το λέμε αυτό διαρροή άνθρακα ή διαρροή θέσεων απασχόλησης ή βιομηχανική διαρροή. Εσείς από τη δική σας προοπτική, γιατί είναι πρόβλημα για την Ένωση πώς θα παραμείνει πρωτοπόρος στην πρόθεση των μέτρων για την ε, κλιματική αλλαγή και χωρίς να χάσει και τη βιομηχανία της. Εσείς από τη δική σας προοπτική πώς το βλέπετε. Είναι πολύ δύσκολο. Ίσως να σας εκπλήσει η ερώτησή μου. Αλλά εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο εύκολες ερωτήσεις δεν υπάρχουν, ούτε εύκολες απαντήσεις. Uh, it's all, if I may ask Andrea for answer. Να, ζητήσω πρώτα, να ρωτήσω πρώτα τον Ανδρέα. Παρακαλώ, πιο σύντομα από ό,τι την πρώτη φορά να απαντήσετε. Ε, Ευχαριστώ. Μάλλον θα μιλήσω αγγλικά γιατί στα γαλλικά δεν τα καταφέρνω καλά. Κύριε Μαρτέν, όταν λέμε ότι θέλουμε κοινότητα για την ε, βιομηχανία, για την για την ενέργεια, τα προβλήματα ε, είναι πιο πολύ στη συμβατότητα. Όταν τα κράτη, τα κράτη-μέλη αναπτύσσουν το καθένα χωριστά την τεχνολογία. Και μετά θέλει το ένα κράτος να καλύτερο από το άλλο και ούτω καθεξής. Άρα είναι μάλλον πολιτικό το πρόβλημα γιατί τεχνικά δεν είναι δύσκολο να λειτουργήσουν τα πράγματα καλά. Αλλά πρέπει να συνεργαστούν οι άνθρωποι. Ιδιαίτερα στην κατάσταση αυτή όπου εμπλεκόνται και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις, μόνο η ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορεί να βελτιώσει τις προδιαγραφές και να αναπτύξει μία ενιαία γλώσσα, ώστε κάθε ψηφιακό μηχάνημα να συνομιλεί με τα άλλα, γιατί μπορούν να συνομιλούν πραγματικά, αλλά πρέπει να ξέρουν την ίδια γλώσσα ή να έχουν μεταφραστές, ιδάλλως δεν μπορούν να επικοινωνούν. Η πολιτική θα το κάνει αυτό. η τεχνολογία, η καινοτομία υπάρχουν. Αλλά πρέπει να αξιοποιηθούν επαρκώς, ευρέως. Και αυτό δεν σημαίνει ε, νέες επενδύσεις τεχνολογία, αλλά μόνο τρόπους για να συνενωθούν οι τεχνολογίες και οι χώρες. Δεν λέμε ότι θα συγχωνεύσουμε την ε, Γερμανία με την ε, Ιταλία ή τη Γαλλία, αλλά δείτε το σαν να μιλάμε για επικοινωνία μεταξύ Ρώμης και Μιλάνου. Ε, και το Παλέρμο βεβαίως. πολύ ωραίο θα ήταν και αυτό. Καλώς, ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Για τον κύριο Μαρτά. Καλό θα ήταν να βρούμε μια τεχνολογία ε, την οποία να μπορούσε να ανθέξει και το βαλάντιο των λιγότερο ευνοημένων στρωμάτων για να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν. Αυτό σημαίνει μια προσέγγιση από τη βάση και για την καινοτομία και για την έρευνα, για τη διαρροή θέσεων εργασίας. Εάν φεύγουν ε, επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Συλλόγω των Θέσεων, για το περιβάλλον και την προστασία του περιβάλλοντος της Ευρώπη, αλλά θέλουν να έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να το αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί δεν μπορεί κανείς βέβαια να φεύγει επειδή αρνείται να δείξει ελληνική με την Ένωση και από την άλλη να ωφελείται από τις αγορές. Νομίζω ότι η λύση πρέπει να είναι αυτή αλλά με το να παίζουν με φόρους ή άλλες νομοθεσίες Νομίζω ότι ένας κατάλληλος ε, φόρος και νομοθεσία τέτοια μπορεί να αποθαρρύνει μια χώρα και αυτό μπορεί να προχωρήσει ε, μαζί με τη λυπή απάντηση για την προστασία του, από την κλιματική αλλαγή, τα χημικά κτλ. Εξαιρετικές οι απαντήσεις σας, ευχαριστούμε πολλά συγχαρητήρια στους νεαρούς φίλους. Ελπίζουμε σε μια άλλη συνεδρία στο Στρασβούργο το Μάιο του 2017, να σας ξαναδούμε, Μάιο του 2017, με, το νέο, με τη νέα συνάντηση του Κοινοβουλίου των Νέων. Χαρήκαμε πολύ που σας είδαμε εδώ, μιλήσατε ανοιχτά, καθαρά και κάτι ακόμη, σημαντική πληροφορία πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, εκ μέρους της Επιτροπής Ήτρες στο Συνολάου της θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία του κύριου Ρίντσε Φανάρουμ, ο οποίος συνταξιοδοτείται ύστερα από μια μακρά και εγκεκριμένη σταδιοδρομία στο, στην Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως στην Ήτρε. Παρακαλώ να σηκωθείτε όρθιος για να σας βλέπουμε όλοι και να σας ε, χαιρετήσουμε. Καλέ φίλε, Ευχαριστούμε πολύ και αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να πω σε όλους εσάς τους νεαρούς ότι σας περιμένουμε γιατί από καιρού καιρών όλο και κάποιος από εμά αναγκάζεται να συνταξιοδοτηθεί και έτσι ανοίγει μια θέση για σας. Είσαστε τόσο καλά προετοιμασμένοι, μιλάτε τόσο ανοιχτά και έτσι ένα λαμπρό μέλλον σας περιμένει, να είστε βέβαιοι. Ευχαριστώ. Great. Και πάω στο σημείο 13. σπουδαίο νούμερο το 13. Ο κύριος Γιώχαν Ντίτριχ Βάνα, Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, όπως ασφαλώς γνωρίζετε πολύ καλά και επιτρέψτε μου γενικέ διευθυντά να σας καλέσω να λάβετε θέση εδώ στο Προεδρείο. Όπως γνωρίζετε, έχει δημοσιεύσει την στρατηγική για το διάστημα της Ευρώπης. Μια νέα στρατηγική, λοιπόν, τον Οκτώβριο δημοσιεύτηκε με πολλά σημεία κρίσιμης σημασίας για αυτή τη ε, βιομηχανία μας, γιατί η καλύτερη πολιτική σημαίνει επίσης, ε, μάλλον πολιτική διαστημική σημαίνει και διαστημική βιομηχανία. Γαλιλαίος, Σπούτνικ, Κοπέρνικος, πώς να βελτιώσουμε την ε, βιομηχανία μας, πώς να την οθήσουμε και είχαμε και την Επίτροπο Βιενκόφσκα, η οποία μας παρουσίασε τη στρατηγική αυτή σε μια προηγούμενη συνεδρίαση, όπου μάλιστα κάναμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα δημόσια ακρόαση. Και η Επιτροπή αρχίσει να εργάζεται για μια έκθεση ίδια πρωτοβουλία για την στρατηγική την διαστημική. Η κυρία Κρέλ, που είναι σήμερα εδώ, θα είναι η συγγήτρια. Είναι η συγγήτρια και ο κ. Ζόρμαρ είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής ε, Διαστημικής, Διαστημικού Οργανισμού, είναι ε, ασχολείται και με το πρόγραμμα Γαλιλαίο και με το Κοπέρνικο. Κύριε Γενικέ, μήπως θα μπορούσατε να πείτε δύο λόγια για τον οργανισμό, γιατί για μένα είναι κάπως νέο αυτό το θέμα. Είναι ένα πεδίο ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ήτρε που είναι σχετικά καινούριο και είμαστε, αισθανόμαστε τεράστια ευθύνη γι' αυτό ακόμα και αν και παλιότερα ήταν στο χαρτοφυλάκιό μας, αλλά δεν είχαμε συγκεκριμένη στρατηγική και δεν είχε εκφραστεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μας ενδιαφέρει λοιπόν πολύ να ορίσουμε το ρόλο σας ως Ευρωπαϊκού Οργανισμού τι δικέ μα εθνικού οργανισμούς και καθώ και όλε τι δραστηριότητε και τι μελλοντικέ δραστηριότητε για το πώ βλέπετε την γενική στρατηγική που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θέλουμε να γίνει συζήτηση για το θέμα. Και να επαναλάβω ότι αισθανόμαστε υπεύθυνοι για το τι συμβαίνει στο διάστημα, αλλά είμαστε υπεύθυνοι και για τα όσα γίνονται στα κράτη-μέλη μας, στη βιομηχανία μας και θέλουμε να βελτιώσουμε τις βιομηχανικές μας δυνατότητες χάρη και στην διαστημική πολιτική. Και η συνεδρίασή μας, κύριε Γενικέ, ε, αναμεταδίδεται ζωντανά στο ίντερνετ, στο νηστότοπο της Επιτροπής Ήτρε, ε, να, την, να βρει τη σημερινή συζήτηση κανείς και στο μέλλον. Και τα επόμενα 100 χρόνια, ίσως. Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα για κανένα μήνα ή από ένα χρόνο μπορείτε να βρείτε αυτή την ε, αναμετάδοση και μαγνητοσκοπημένη. Και γι' αυτό σας δίνω αμέσως το λόγο, κύριε Γενικέ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω με την ευκαιρία αυτή της συζήτησης για το τι μπορούμε να προβλέψουμε για το μέλλον. Θα προσπαθήσω να ε, ανταποκριθώ ακριβώ στο αίτημά σας, κύριε Πρόεδρε, να σας εξηγήσω τι κάνει η ΕΖΑ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και τι νόημα έχει αυτή η στρατηγική της Επιτροπής για μας. Ε, θα δείτε ότι όλα αυτά θα τα συνενώσω, ελπίζω ότι θα μπορέσω ε, έτσι ώστε να καταστεί σαφές το νόημά μου. Να κοιτάξουμε λοιπόν τι έχουμε ήδη. Είχαμε τον αγώνα για το διάστημα ε, με ακριβώς αυτό το θέμα. Ε, Ποιο δηλαδή θα είναι ο πρώτο που θα στείλει τον άνθρωπο στο διάστημα και το σχετικό κύρο που αυτό συνεπαγόταν ε, για, για τι υπερδυνάμει τη ΗΠΑ, Ρωσία, την ιστορία την γνωρίζετε ασφαλώ, πώ κατέληξε αυτό το τόσο ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπορώ να πω ότι ή μη τι άλλο Είχε λεφτά το διάστημα τότε, ρίχναμε λεφτά στο διάστημα, ήταν το μόνο θετικό, τα λοιπά όχι και τόσο. Τώρα η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική, τελείως διαφορετική θα έλεγα. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε το διάστημα, μπορεί να γεφυρώσει κρίσει επίγειες. Η κρίση της Κρυμαίας βεβαίως το γνωρίζουμε και θα πρέπει να έχει ο καθένας τη δική του πολιτική θέση και στάση, αλλά ταυτόχρονα στέλνουμε αυστροναστροναύτες από την Ευρώπη, από τις ΗΠΑ, από τη Ρωσία, από τον Καναδά, την Ιαπωνία, μέσα σε μια μικρή κάψουλα στον ε, Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, χωρίς να του ζητάμε θεώρηση διαβατηρίου. Και είναι πολύ καλό, πολύ θετικό το ότι μπορούν ακόμη και κατά τη διάρκεια επιγείων κρίσεων που είναι να εξελίξει να συνεργάζονται αυτοί εκεί. Βεβαίω θα υπάρχουν και κάποιε πολιτικέ δράσει, το γνωρίζω αυτό, αλλά ελπίζω ότι τουλάχιστον μετά την, ε, μετά την εκδήλωση των κρίσεων να μπορούμε να τα γεφυρώνουμε αυτά. Ξέρετε ποιες είναι οι παγκόσμιες προκλήσεις. Ε, έχετε την δική σας ε, προοπτική για τις παγκόσμιες προκλήσεις. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε τον κατάλογο. Ναι, τον βλέπετε. Δεν ξέρω αν μπορείτε να διαβάσετε τα γράμματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε μια εικόνα, έναν αρκετά εξαντλητικό κατάλογο. Κλιματικές αλλαγές, μετανάστευση, κινητικότητα, επικοινωνία, ε, ενέργεια και... Και βλέπετε τελευταία γραμμή αυτό το παράξενο που δεν είναι μια πρόκληση ή κρίση, αλλά ε, είναι ο κινητήριος μοχλός που κινεί την γη, η περιέργεια. Είναι η περιέργεια αυτή που μας έκανε να αφήσουμε τη σπηλιά ε, και να προχωρήσουμε και μας έχει κάνει να ταξιδέψουμε πέρα από τα όρια των ε, υπήρων μας. Είναι μεγάλο κίνητρο λοιπόν η περιέργεια. Η Ευρώπη πάντοτε χαρακτηριζόταν από αυτόν τον μεγάλο κινητήριο μοχλό την περιέργεια, όχι μόνο με τον Κολόμβο και με πολλούς άλλους εξερευνητές. Τα παιδιά, τα παιδιά που έχουν αυτή τη φυσική περιέργεια και που κοιτούν δεξιά-αριστερά, που δοκιμάζουν κάτι διαφορετικό και που βλέπουμε τους γονείς τους να είναι τόσο υπερήφανοι. Αν είχαμε την ίδια περιέργεια λοιπόν και ως ε, πιο ηλικιωμένοι, και δεν λέω να δοκιμάζουμε μια διαφορετική γεύση, ένα φαγητό, θα είχε πάρα πολύ μεγάλα, μεγάλη σημασία ένας καθηγητής όπως εγώ ας πούμε να δοκιμάζει να αναζητεί κάτι καινούριο. Η περιέργεια λοιπόν μας φέρνει στο διάστημα, στη πληροφορία μπορούμε να αντλήσουμε από τους δορυφόρους, κλιματικές αλλαγές, μετεωρολογικές συνθήκες κτλ. Αλλά και σε επικοινωνία αλληλεπίδραση στην Ευρώπη μεταξύ διαφορετικών πολιτικών συστημάτων, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στην Ευρώπη, και μπορούμε και να εμπνεύσουμε με τους νέους στο δρόμο για το μέλλον, γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι πτυχές, τρομοκρατικές επιθέσεις, κλιματικές αλλαγές, οικονομική κρίση. Υπάρχουν προβλήματα πολλά. Πρέπει όμως να τους δείξουμε και ότι αξίζει τον κόπο να δουλέψουν για το μέλλον, για ένα μέλλον καλύτερο. Και το μέλλον να βλέπετε όπως και στο παρελθόν. Να, οι δεινόσαυροι με τη γελιογραφία που βλέπετε παρακολουθούν ένα μετεωρίτη να πέφτει. Ξέρετε ότι μετεωρείται σήμερα το τέλος των ε, δεινοσαύρων. Δεν αρκεί λοιπόν κανείς να διατυπώνει μια ευχή. Πρέπει να πράττει κιόλα και αυτή είναι η δική μας προσέγγιση. Μιλήσαμε για διαφορετικά κίνητρα. Όπως είπα, το κίνητρο του κύρους ήταν αυτό που κινούσε τις μεγάλες δυνάμεις κατά τον ψυχρό πόλεμο. Ωστόσο, έχουμε τώρα διαφορετικά κίνητρα, ε, άλλες επιχειρήσεις, δυτικό φορέα κτλ. Έχουμε διαφορετικούς ε, παράγοντες που δραστηριοποιούνται στο διάστημα και μάλιστα και έτοιμα από διαφορετικές πηγές ε, που διαθέτουν και χρήμα για να αναπτυχθούν άλλες δραστηριότητες στο διάστημα και πια το περιεχόμενο έχει αλλάξει σχέση με το διάστημα. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει μόνο να στείλουμε τον άνθρωπο στο διάστημα αλλά να κοιτάξουμε τις λεπικοινωνίες, την πλοήγηση, ε, και βέβαια έχει αλλάξει και το σύνολο των ρόλων που διαδραματίζει ο καθένα. Οι υπηρεσίε στο μέλλον δεν θα είναι μόνο υπηρεσίε που θα ανοίγουν πορτοφόλι και θα πληρώνουν, αλλά θα έχουν τελείω διαφορετικό ρόλο και θα περάσω αυτό μετά. Αλλάζει βέβαια και το σύνολο των τεχνολογιών. Εσεί μιλήσατε νωρίτερα για την ψηφιοποίηση, η οποία τώρα ξεπερνάει τα όρια τα γήινα και περνάει στο διάστημα με έναν εκτοξευθεί τρισδιάστατο, με, ηλεκτρονική, με τρισδιάστατη εκτύπωση που μπορεί να παραχθεί και άρα περνάμε σε μια νέα εποχή του διαστήματος. Κάποιοι λένε νέο διάστημα. Για μένα δεν αρκεί αυτό. Για το νέο διάστημα σημαίνει εμπορευματοποίηση. Εμπορευματοποίηση του διαστήματος γίνεται και στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αλλά μιλούμε για μια νέα ιδέα του διαστήματος και την εμπορευματοποίηση και την ε, πληροφορία στον πολίτη, την ενημέρωση, την έμπνευση, τις θέσεις εργασίας, την ψηφία την ε, αλληλεπίδραση. Ένας νέος λοιπόν όρος για, ε, για το διάστημα. Η ΕΖΑ λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, έχει ρόλο να συνενώσει όλους αυτούς τους παράγοντες, την πολιτική, την κοινωνία, την επιστήμη και την βιομηχανική παραγωγή. Όλα αυτά είναι το Space 4.0. Ε, με τη συζήτηση που αναπτύξαμε μεταξύ των 22 μελών μας, που είναι παράλληλα στο μεγαλύτερό του βαθμό και μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν τη Ελβετία και τη Νορβηγία και του συνδεδεμένου μέλου που είναι η Σλοβενία και του Καναδά που συνεργάζεται μαζί μας, αλλά και τα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν συμβατικές σχέσεις μαζί μας και έχουν ζητήσει τη συνεργασία. Με όλους αυτούς λοιπόν τους φορείς κάναμε συζήτηση πολιτών μέσα σε μία μέρα, ένα Σάββατο, με 2.000 συμμετέχοντε σε διαφορετικά κράτη-μέλη, όπου συζητήθηκε τι είναι το διάστημα, σε τι μας χρησιμεύει, τι να κάνουμε στο μέλλον, τι θέλουμε να βλέπουμε στο μέλλον για το διάστημα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση σε ηλικίε 15 ε, έως 89, βλέπετε και ηλικιωμένους λοιπόν, πολύ ηλικιωμένους στην εικόνα μας, αλλά και πολύ νέους. Ε, φοβερά ενδιαφέρουσα η συζήτηση, δεν μπορώ να σας λεπτομερή αποτελέσματα, αλλά τα έχουμε στην ε, σελίδα μας λεπτομερώς, πάντως προκύπτει κάτι ξεκάθαρο. Πρώτον ότι υπάρχει σαφέστατη εμπιστοσύνη, πολύ καλά τα ποσοστά και αυτό μας ενθαρρύνει, στην υπηρεσία μας και γενικά τις υπηρεσίες διαστήματος και φτάνω στο τέλος της διαφάνειας αυτής όπου βλέπουμε κατά 81% ο κόσμος να ζητάει να εκμεταλλευτούμε τους φυσικούς σπόρους του διαστήματος. Εγώ το πολύ πολύ 20% είναι υπολόγιζα, αλλά όμως το 80% και άνω μας λέει να αξιοποιήσουμε τους σπόρους του διαστήματος, αλλά ταυτόχρονα μας λένε προσοχή, μην καταστρέψετε το διάστημα, μην ρυπάνετε το διάστημα. Αυτά λοιπόν έχουν τεράστια σημασία, αποτελούν ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα και ο κόσμος, ο κόσμος που δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Έχουμε πολλά ε, και ποικίλα κράτη-μέλη και κράτη γενικότερα στην Ευρώπη. Η ΕΖΑ λοιπόν ως εκ της φύσεως της και καθώς έχει ήδη 22 ε, μέλη κράτη ε, ε, και, και κράτη Ευρώπης μαζί με τον Καναδά έχει ήδη ε, προσέγγιση για το πώς μπορεί να δράσει στο παγκόσμιο σκηνικό. Έχουμε μέλη από διάφορες εθνικότητες, όχι μόνο Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για συνεργασία, για διαμεσολάβηση, για διευκόλυνση και συμμετοχή Φερρυπίν και της βιομηχανίας στην πορεία αυτή στο διάστημα. για την καινοτομία που ρωτήσατε. Πρέπει να την προσδιορίσουμε καταρχά την καινοτομία. Για μένα η καινοτομία είναι το να μπει μια, ένα προϊόν στην αγορά. Η καινοτομία δεν είναι μόνο μια νέα ιδέα, όσο και αν πολλέ φορέ με, με αυτήν την έννοια χρησιμοποιείται ο όρο, αλλά η καινοτομία για μένα είναι να μπει το προϊόν στην αγορά. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε την αλυσίδα τη καινοτομία από την πολύ βασική έρευνα μέχρι και την ε, κυκλοφορία στην αγορά ενό προϊόντο. Αυτή είναι η αλυσίδα την οποία με πολύ μεγάλη προσοχή ε, ε, προωθεί η ΕΖΑ, να μην υπάρξει αυτή η λεγόμενη κοιλάδα του θανάτου, να μην υπάρξει η ρήξη δηλαδή των κρίκων. Και φυσικά αυτό το κάνουμε μόνοι μα, αλλά θέλουμε από τη βασική έρευνα να φτάσουμε μέχρι τη διάθεση στην αγορά του προϊόντο. Αυτό σε συνεργασία πάντα με πανεπιστήμια, με ερευνητικά κέντρα κτλ. Και όπω είπαμε, αυτό αλλάζει το, το, το, το διάστημα. Το διάστημα 4-0 όλο και περισσότεροι είναι οι φορεί και οι, ε, τα πρόσωπα, τα νομικά που μπαίνουν σε αυτήν την προσπάθεια για την παραγωγή προϊόντων συγκεκριμένα που ενδιαφέρουν τον καταναλωτή και για την καινοτομία. Ε, βεβαίως μπορεί να γίνει καινοτομία για τη χρήση στο διάστημα, για μετά να εφαρμοστεί στην αυτοκινητοβιομηχανία, σε διάφορους άλλους τομείς. Όρια δεν υπάρχουν. Αυτή είναι μια λύση βέβαια. Και η Ευρώπη έχει μια τεράστια ευκαιρία μια τεράστια ευκαιρία αυτή η αλυσίδα της ε, καινοτομίας να αναπτυχθεί περισσότερο και ιδιαίτερα γιατί παραδείγματι δεν υπάρχουν ε, τρόποι υπολογισμού της κατανομής ε, του της αστικής συγχωρήπανσης από το διάστημα. Γιατί να μην υπάρχει αυτός ο μηχανισμός υπολογισμού, μέτρησης καλύτερα, της αστικής συγχωρήπανσης από το διάστημα και επίσης θα πρέπει να υπάρχει και ένας στενός συσχετισμός μεταξύ διαστήματος και άλλων τομέων. Αυτό κινήτων παραδείγματι που μέσα από την αλυσίδα αυτή μας επιτρέπουν ένα αυτόνομο δίκτυο, δηλαδή μπορούμε το διάστημα να το αξιοποιούμε ε, για τόσα πράγματα πάνω στη γη. Ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι ανοιχνευτές πυρκαγιάς που έχετε εδώ μέσα στην αίθουσά σας υπάρχουν επειδή έπιασε φωτιά το Απόλλων 1. Επειδή έπιασε φωτιά το Απόλλων 1 δημιουργήθηκε ο ανοιχνευτής πυρκαγιάς, ο ανοιχνευτής καπνού. Τόσες πολλές είναι οι δημιουργικές δυνατότητες που μας προσφέρει το διάστημα. Ε, υπάρχουν τα κέντρα επίσης... Ε, θερμοκοιτίδων θα λέγαμε του διαστήματος, εκεί δηλαδή όπου δίνουμε ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες αλλά και σε πιο ηλικιωμένους εφόσον έχουν τη δυνατότητα της καινοτομίας να ανοίξουν ε, νέες δυνατότητες με νέες θέσεις και θέσεις εργασίας βεβαίως. Ε, θα έχετε ακούσει για να σας δώσω ένα παράδειγμα να γίνεται λόγος για τη Ροζέτα με τον Γερασιμένκο. Επιστήμη. 100% επιστήμη. Βλέπετε όμως, ένας κομίτης σκούρος, μαύρος, σαν το, σαν το κάρβουνο, και πάει η ροζέτα με μία ε, κάμερα που ξεχωρίζει το σκούρο γκρι από το πιο ανοιχτό γκρι, το ενδιάμεσο κτλ. Και τώρα, μετά τη δημιουργία αυτής της εφεύρεσης, μπορεί να πάει στο δάσος, η ίδια κάμερα, να πετάξει πάνω από ένα δάσος και να κοιτάξει αν υπάρχει κάποιο ίχνος γκρι που μπορεί να είναι ένα τηγάνι τεφάλ. Μην, πω, μην ξεχάσω να πω ότι και το τεφάλ, το τεφλόν δηλαδή προέρχεται από την διαστημική έρευνα ή να είναι καπνός φερρυπίν ε, που μπορεί να είναι επικίνδυνος για πυρκαγιά στα δάση. Αυτά λοιπόν, εγώ προσωπικώς ε, έμαθα ότι πρέπει το ευρωπαϊκό πνεύμα να μείνει και για το μέλλον. Οι γονεί μου με δίδαξαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να οδηγήσει στις ευρωπαϊκές πολιτείες, στις ενωμένες ευρωπαϊκές πολιτείες. Αυτό ίσως είναι μια συζήτηση για το μέλλον. Αλλά εδώ βλέπετε το πραγματικό πνεύμα του μέλλοντος. Η γαλλική τηλεόραση, δεν είναι εδώ ο Γάλλος βουλευτής πια, αλλά μου αρέσει πολύ αυτή η εικόνα γιατί βλέπουμε τη γαλλική τηλεόραση και στα δεξιά σας ο αστροναύτης δεν είναι Γάλλος, είναι Ευρωπαίος αστροναύτης Βρετανικής εθνικότητας. Επί 20 λεπτά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ε, έδωσε συνέντευξη από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Να λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε και από το διάστημα να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό πνεύμα συνεργασίας. Είναι κάτι το οποίο για μένα σημαίνει πως από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μας οδηγήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης. Μπορεί να μην είναι για το άμεσο μέλλον, αλλά εγώ μπορώ να προσπαθήσω, μπορώ να υποστηρίξω και μπορώ να βοηθήσω στη δημιουργία του Ηνωμένου Διαστήματος για την Ευρώπη, γιατί έχουμε φορείς πολύ ισχυρούς και ιδιαίτερα κρατικού ε, του κρατικού τομέα, του δημόσιου τομέα και από τα κράτη και από την ΕΖΑ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συνεργασία τους και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Η σύμβαση της ΕΖΑ ανάγεται στο 1975. Έκτοτε έχει η ΕΖΑ αναπτύξει μια σειρά από τομείς δραστηριοτήτων. Βλέπετε ένα καλλιδοσκόπιο εδώ της δράσης μας, ε, πλοήγηση, τηλεπικοινωνίες, επιστήμη του διαστήματος, ε, διερεύνηση, νέα συστήματα εκτόξευσης ε, διαστημικά, οχήματα, επανεισόδου, ε, δράση στο διάστημα, προφύλαξη της γης ακόμη σε περίπτωση κινδύνου από μετεωρίτη, πρέπει να έχουμε τα μέσα αυτά για να προφυλαχθούμε για το μέλλον. Αν τυχόν έχει δει κάποιο από εσά την ταινία Αρμαγεδόν, πιστεύω θα έχει πιστεί πω χρειαζόμαστε τα δικά μα μέσα για την προστασία από ενδεχόμενου μετεωρίτε. Ε, έχουμε λοιπόν την ΕΖΑ ε, που υποστηρίζει μαζί με τα κράτη-μέλη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο τις μεγάλες, τους μεγάλους ομίλους και τις συμπράξεις. Και μετά έρχεται η συνθήκη της Λισαβόνας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτή η συνθήκη της Λισαβόνας Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να πάψει να υπάρχει ΕΖΑ, αλλά υπάρχει μια σαφέστατη φράση τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Είναι μικρά τα γράμματα και δεν μπορείτε να τη διαβάσετε, αλλά σα το διαβάζω εγώ. Λέει ότι πρέπει να υπάρχουν καλέ σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΕΖΑ. Αυτό λοιπόν το οποίο διαβάζουμε τώρα, αυτό που ακούμε τώρα με την κυρία Σβιατκόφσκα για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική του Διαστήματος, για να δούμε πού εγγράφεται εδώ, γιατί προσπαθούμε να το τοποθετήσουμε με αυτή την εικόνα. Υπάρχουν κοινή ευρωπαϊκή στόχη ασφαλώς, συνοχή, κοινό ευρωπαϊκό πνεύμα κτλ. Υπάρχει επίσης η κοινή διακήρυξη ΕΖΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπεγράφει από τον υποφαινόμενο και την κυρία Βιενκόφσκα και ορίζει τους ε, γενικούς στόχους ε, ενσωμάτωση του διαστήματος στην καθημερινή ζωή, ένωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, ευρωπαϊκή αυτονομία στρατηγική σημασία τομής ε, και βέβαια το, η συμφωνία πλαίσιο που τα περιγράφει όλα αυτά. Άρα εδώ βλέπετε ευρωπαϊκό πνεύμα συνοχή και κάτω από αυτό, από την κοινή διακήρυξη, τους ε, ειδικού στόχους που αναπτύσσουν η ΕΖΑ αφενός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αφετέρου. Μιλήσατε εσείς για την στρατηγική για το διάστημα της Επιτροπής, στρατηγική για το διάστημα, νέοι στόχοι, αφενός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφετέρου η ΕΖΑ, και πιστεύω ότι θα επικυρωθούν ε, γιατί έχουμε στην Λουκέρνη μία ε, υπουργική συνεδρίαση των ε, υπουργών που εκπροσωπούν όλα τα κράτη-μέλη, ε, διάστημα 4.0. Στη Λουκέρνη, όπως σας είπα, και περιμένουμε να επικυρώσουν αυτές τις δηλώσεις με την κοινή τους διακήρυξη, που θα αποτελέσει μια πολύ καλή έμπνευση για το μέλλον. Να σε εργαστούμε λοιπόν όλοι μαζί για το μέλλον, γιατί έξω από την Ευρώπη είναι ανταγωνιστές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε έτσι μια εμπνευσμένη ομιλία τώρα που ξεκινάμε τις δραστηριότητε μας στο θέμα αυτό. Εκ μέρους του ΕΛΚ τώρα, η κυρία Γκροστέτ, αντιπρόεδρος. Παρακαλώ. Κύριε Διευθυντά, καταρχήν σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας. Όχι μόνο η παρουσία σας ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αλλά ήταν και ενθουσιώδης. Ε, πραγματικά μεταδώσατε τον ενθουσιασμό σας. Ε, ε, αντιλαμβανόμαστε έτσι όλα αυτά αυτά που πρέπει να ε, τοποθετήσουμε σε αυτή τη στρατηγική και πώς η Ευρώπη μπορεί εδώ να συσπυρώσει και συμφωνώ ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτά που είπατε. Ε, η υπηρεσία του διαστήματος άλλωστε ε, είναι σε μια καλή περίοδο, επιβεβαιώθηκε το Αριάν 6, είχαμε την επιτυχή εκτόξευση 5 δορυφόρων Γαλιλαίο από το Αριάν 5 στο, ε, διαστημικό σταθμό όλα αυτά ε, όλες αυτές επιτυχίες έχουν να κάνουν με μια ε, σημαντική ευρωπαϊκή εμπλοκή και πρέπει να συνεχίσουμε να εμπλεκόμαστε και να δεσμευόμαστε και μέσω των προπολογισμών μας, ε, αλλά και μέσω της εμπιστοσύνης που δείχνουμε ε, στην Ένωση, στην υπηρεσία σας είναι σημαντικό για την εξαρτησία της Ευρώπης. Ξέρουμε ότι η Ήπειρός μας πρέπει να είναι ανεξάρτητη και στον τομέα του διαστήματος. Γι' αυτό λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε μια πραγματική πολιτική, βιομηχανική πολιτική στον τομέα του διαστήματος. Ε, είναι στρατηγική σημασίας. Τα μεγάλα προγράμματα Κοπέρνικος, Γαλιλαίο, πλέον ε, παίρνουν σάρκα και οστά και πρέπει να ε, στηριχτούν. Ε, είναι σημαντικές επιπτώσεις για όλους. Ε. Το είπατε και στην παρουσίασή σας. Οι συμπολίτες μας πρέπει να οικειοποιηθούν αυτήν την ευρωπαϊκή πολιτική διαστήματος. Είναι σημαντικό για την προστασία των συνόρων, για την προστασία του περιβάλλοντος, τον τομέα της αεροναυπηγικής, της ε, ιατρικής και άλλους πολλούς τομείς. Όλα αυτά τα δεδομένα ε, πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε καλύτερα. Αυτή είναι η δουλειά που έχουμε σήμερα. Σε σχέση τώρα με τον περίπλοκο χαρακτήρα υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, ε, ποιες είναι οι βελτιώσεις που η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία μπορεί να επιφέρει ε, στον τρόπο με τον οποίο συντονίζει και διαχειρίζεται τα προγράμματα αυτά από κοινού με τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι δεν είναι πάντα εύκολο, εύκολος ο συντονισμός. Μας παρουσιάσατε έτσι μια εικόνα, εντάξει όχι ιδηλιακή, αλλά εξαιρετικά ενθουσιώδης. Θα πρέπει να υπάρχουν και δυσκολίες. Ποιες είναι αυτές τις δυσκολίες λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πώς θέλετε να σας βοηθήσει. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια ορατότητα της δράσης μας στον τομέα του διαστήματος. Να είναι σαφές ε, και προφανές για όλους. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών η κυρία Κρέλ, η οποία είναι και η συγγήτρια για το σύνολο της Επιτροπής Ήτρε. Ναι, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ κύριε Βερνάρ για την πολύ ενθουσιώδη αυτή η παρέμβαση. Ελπίζω να μας άκουσαν και πολλοί από το ίντερνετ γιατί είναι συναρπαστικά αυτά που μας είπατε. Όπως έχει μάλιστα το γενικό κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω ότι ήταν και πολύ χρήσιμη η δική σας παρέμβαση. Όπως ε, ακούσατε είμαι η συγγήτρια για την έκθεση πρωτοβουλία στρατηγική για το διάστημα. Υπολογίζω κάπου το Μάρτιο να καταθέσω στην Επιτροπή μας την ε, πρόταση. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι παρούσα στην ακρόαση γιατί έλειπα από τις Βρυξέλλες εκείνες τις μέρες. Είχα την ευκαιρία όμως την ίδια εποχή στην Χιλή να πάω να δω το ε, Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Διαστήματος ένα καταπληκτικό παράδειγμα της ευρωπαϊκής συνεργασίας με αποτελέσματα απτά και συναρπαστικό είναι να βλέπει κανείς ότι επιστήμονες, άντρες και γυναίκες, δυστυχώς περισσότεροι άντρες παρά γυναίκες, είναι εκεί για να συνεργάζονται, προέρχονται από όλη την Ευρώπη με καταπληκτικά αποτελέσματα και επίσης Ένα ζήτημα που έχει να κάνει και αφορά βέβαια και τη στρατηγική μας ήταν αυτό της επικάλυψης συχνοτήτων που έχει μεγάλη σημασία και για τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ίσως περιλάβω κάτι στην έκθεσή μου, αν μου δώσετε και σας καποιο εναυσμα έναρσμα. Ένα-δύο ζητήματα θα ήθελα να ε, σημειώσω κατόπιν ε, της για να ακούσω μετά και τι γνώμη έχετε Φιρυπίν τι μέτρα βλέπετε ε, να απαιτούνται σε σχέση με την προσέγγιση στην αγορά. Οι προτάσεις Επιτροπής Αρχού, αρκούν, πρέπει να έχουμε μια πιο ε, επίμονη προσέγγιση. Επίσης, η ιδιωτική αγορά έχει ασφαλώς τεράστια σημασία στην δευτερογενή αξιοποίηση της ε, τεχνολογίας, αλλά πιστεύετε ότι και για την πρωτογενή ε, παροχή των υπηρεσιών πρέπει να είναι παρούσα η ιδιωτική αγορά. Ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο έχει δοκιμαστεί στις ΗΠΑ, αλλά ήταν πολύ μέτρια τα αποτελέσματα. Δεν ε, ξέρω εάν έχει ιδιαίτερη σημασία να κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια. Εσείς τι πιστεύετε. Για μένα μεγάλη σημασία θα έχει ιδιαίτερα μη στρατιωτικού χαρακτήρα ε, εγχειρήματα για το διάστημα να παίρνουν την πρωτοπορία. Φυσικά δεν θα λησμονήσουμε την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι ε, αμεληταίο ζήτημα, αλλά η μη στρατιωτική φύση των προγραμμάτων πιστεύω ότι θα πρέπει να παίρνει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο από αυτό το κομμάτι, από τα προγράμματα. Ε, και επίσης, διαστημικά απόβλητα και ρήπανση του διαστήματος έχουν κεντρική και όλο και πιο κεντρική σημασία λαμβάνουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει κάποιες προτάσεις με τη νέα στρατηγική, αλλά και εδώ πιστεύω η ΕΖΑ θα έχει τεράστιο ρόλο να διαδραματίσει. Ο προπολογισμό που έχετε στη διάθεσή ή που θα έπρεπε να έχετε στη διάθεσή Πώς προχωράει, έχει διευκρινιστεί αυτή, έχει διευκρινιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί ίσως θα πρέπει και εμείς αυτό να το περιλάβουμε στην γνωμοδότησή μας και στην έκθεσή μας και επίσης προσθέτως αυτόν που είπε η Επιτροπή με το σχεδιασμό της. Τι άλλο πιστεύετε ότι είναι σημαντικό και πρέπει να περιλάβουμε στην έκθεσή μας. Ευχαριστώ κύριο Στυζενεύσικη από την ομάδα ECR Ευρωπαίων Στηρητικών Μεταρρυθμιστών. Eh, eh, ευχαριστώ, θα μιλήσω τσέχικα. Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα εισαγωγικά σχόλια όπου και αναφερθήκατε ε, την ε, υπηρεσία διαστήματος και στις επιτυχίες της. Είπατε ότι στο παρελθόν η έρευνα στον τομέα του διαστήματος ε, ε, είχε το κίνητρο του ανταγωνισμού μεταξύ των υπερδυνάμεων. Αναφερθήκατε στην κούρσα προς το διάστημα. αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι το διάστημα είναι ανοιχτό για όλους. Και ουσιαστικά το επιχειρηματικό πνεύμα είναι αυτό που κινεί την έρευνα στο διάστημα. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρυνθούν οι start-up. Το διάστημα είναι μια τεράστια ευκαιρία για νέους ανθρώπους, για καινούργιες εταιρείες. Γενικότερα η έρευνα στον τομέα του διαστήματος ε, αρχίζει να γίνεται μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δραστηριότητα, ένας ενδιαφέρον κλάδος για τις επιχειρήσεις και για την έρευνα. Θέλω να σας συγχαρώ, διότι από ό,τι φαίνεται ε, είναι κάτι το οποίο δεν έχει τονιστεί επαρκώς ε, για την ε, θέση τροχιά των τεσσάρων ε, δορυφόρων Γαλιλαίου. Είναι τεράστιο επίτευγμα τέσσερις δορυφόρες, δορυφόροι συγγνώμη, ταυτόχρονα. Ελπίζω να λειτουργήσουν όλοι καλά και ελπίζω το ερχόμενο έτος τον Γαλιλέω να είναι ανοιχτό για όλους, διότι τότε είναι που θα γίνει πραγματικότητα. Εξού και το ερώτημά μου. Οι νέες ευκαιρίες επιχειρηματικές που δημιουργούνται σε σχέση με το διάστημα είπατε ότι υπογράφηκε μια σύμβαση έρευνας για το Αριάν 6. Αυτό είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο, διότι δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για νέα συστήματα. Ε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, πότε πιστεύετε ότι θα έχουμε νέα συστήματα όπως το Αριάν 6 που να μπορούν να λειτουργήσουν το θέτω το ερώτημα αυτό, διότι ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα θα κινηθούμε και εμείς στις εργασίες μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, διότι πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος έχει πραγματικά σημειώσει τεράστια βήματα προόδου. Είναι μια, ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό επίτευγμα. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα η κόρα Von Χάουζεν. Ευχαριστώ τον κύριο Βέρνερ για την ε, πραγματικά ε, πολύ ζωντανή ε, και ενθουσιώδη παρουσίαση για αυτόν εξαιρετικά θετικό. Χαίρομαι ιδιαίτερα που διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία έχουν υπογράψει μια κοινή δήλωση για, το, για την πολιτική διαστήματος, κατά την παρουσίαση στρατηγικής διαστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι ένα μήνυμα ε, είναι η στιγμή να σπάσουμε τα στεγανά και να συνεργαστούμε. Αυτή η στρατηγική για είναι ένα πλήρες έγγραφο. Μας αρέσει ο γενικότερος τόνος, μεγαλύτερος ρόλος για τον ιδιωτικό τομέα. Θέλουμε τα εμβληματικά μας προγράμματα να αποδώσουν. Ε, η κυρία Γκροστέτ ε, αναφέρθηκε και αυτή στο γεγονός ότι το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει ε, το πώς το διάστημα και οι δραστηριότητες στο διάστημα επηρεάζουν την καθημερινή του ζωή. Οπότε το ίδιο ερώτημα ε, θέλω να θέσω και στην Επίτροπο Μπιανκόφσκα. Θα πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη ε, στρατηγική επικοινωνία, να μην επικεντρωθούμε μόνο στο χωριό, στο διάστημα, έτσι, να μιλήσουμε για βασικά πλεονεκτήματα που μας παρέχει το διάστημα στη καθημερινότητά μας. Είναι ένας πολύ μεγάλος, μεγάλος και σημαντικός κλάδος, όμως ε, με την Πίτρο Μπιανκόφσκα, ε, εγώ, εσείς, ε, νομίζω κάναμε μια προσπάθεια για να εκπροσωπηθούν και οι γυναίκες, διότι είπατε ότι είναι ένας ανδροκρατούμενος κλάδος. Θα πρέπει να υπάρξουν και περισσότερες επενδύσεις όμως διότι αν δεν συνειδητοποιήσουν ε, πόσο σημαντικό είναι για την καθημερινότητά μας ε, ο κλάδος αυτός, τότε είναι πιο επιφυλακτικοί στο να επενδύσουν. Ε, και δύο ακόμα ερωτήματα για τις πλατφόρμες δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική το διάστημα αναφέρεται ε, στο να τη δημιουργία μιας πλατφόρμας διάδοσης στοιχείων για να ε, ενθαρρυνθεί η δυνατότητα του Κοπέρνικου κυρίως. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν πότε αυτές οι πλατφόρμες θα είναι λειτουργικές και ποια είναι τα βασικά κριτήρια για τις προμήθειες, για το διαγωνισμό που θα γίνει. Η διαλειτουργικότητα ε, θα είναι εύκολο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν και να ε, επωφεληθούν τις πλατφόρμες αυτές. Και τελευταίο ερώτημα, Πρόεδρε, για τους ε, μικρούς εκτοξευτές ε, είδαμε ότι έχουμε όλο και πιο μικρούς ε, ε που τίθεται σε τροχιά που είναι πιο εύκολο να, να εκτοξευθούν όμως το Βίγκα μπορεί να εκτοξεύσει μόνο ε, ε, δορυφόρους βάρους 300 κιλών που ξεκινούν από 300 κιλά μπορούν, μπορεί να εκτοξεύσει και πιο μικρούς δορυφόρους υπαρχική δυνατότητα σύμπραξης δημοσίου τομέα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Κόχλιτσεκ. Ε, και ο Κόχλιτσεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η παρουσία σας κύριε Βέρνερ ήταν εξαιρετικά ζωντανή και πιστική. Είναι κρίμα που δεν ξέρει το ευρύ κοινό τι συμβαίνει στον κλάδο αυτόν. Μπορεί κάποιο να μα σταματήσει κάποιο στον δρόμο στο, στο Βέλγιο να το ρωτήσει τι είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο και θα νομίζει ότι του λέω κάτι εξωγήινο. Ε, πρέπει παντού αυτές οι παρουσιάσεις να γίνουν. Το ερώτημά μου λοιπόν το εξής. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει μια διεθνή σύμβαση ε, για την μείωση του μη επιθυμητού υλικού στο διάστημα. Δεν θέλουμε η μόλυνση, ε, να μολύνουμε το διάστημα όπως μολύναμε τη γη. Ε, ένα άλλο ερώτημα τώρα. Τον Γαλιλαίο. Πιστεύετε ότι θα έχετε εκτοξεύσει και στους 30 ε, Δορυφόρου στο προσεχές μέλλον και ποιο είναι λίγο πολύ το χρονοδιάγραμμα. Πότε όλοι αυτοί οι δορυφόροι θα τεθούν στη τροχιά και θα λειτουργούν και αυτοί που είναι ενεργοποιηθούν και οι, οι, οι δορυφόροι υποκατάσταση. Τώρα, η Διεθνής Διαστημική Σταθμή, ξέρετε ότι τελειώνει ο κύκλος ζωή του. Ε, η Ευρώπη θα συμμετάσχει στην ε, οικοδόμηση κάποιου νέου δημοσιονομικού σταθμού. Πώς σκοπεύουμε να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό; Είναι από αυτά τα ελκυστικά θέματα, όπως είπε προηγουμένως και η συνάδελφος. Και το τελευταίο, πώς θα δημοσιοποιείτε τα δεδομένα τα οποία φτάνουν στα χέρια σας. Φαντάζομαι ότι φτάνουν κάποια δεδομένα στα χέρια σας ε, οι παρατηρήσεις ε, των, ε, του ορατού και του μη ορατού φάσματος. Τα δεδομένα αυτά είναι εξαιρετικά χρήσιμα για διάφορες τεχνολογίες. μπορεί να χρησιμοποιηθούν και στον τομέα της αρχαιολογίας, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν λοιπόν τεράστιε δυνατότητε αλλά και ο τομέα τη αλληλεία, της ε, του περιβάλλοντος. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ομιλητές. Ο κύριος Ζωρίνιο τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γενικό για την ε, ωραία εισήγηση που μας έκανε για τη στρατηγική 4.0. Ήταν μια εισήγηση πολύ εμπνευσμένη και η συζήτηση που είχαμε ε, την τελευταία φορά με τους επιτρέπους Εύκοβιτς και Πιενκόφσκι ήταν ιδιαίτερα ε, ενδιαφέρουσα. Πρέπει βέβαια η στρατηγική να έχει σαφείς στόχους, αλλά μετά πρέπει να χρηματοδοτήσει διάφορα project και πρέπει να θεωρηθεί ως μια σφαιρική προσπάθεια με ένα καλύτερο, για έναν καλύτερο κόσμο, ε, ένα καλύτερο πλαίσιο για τη συνεργασία μετά την κρίση. Εγώ θα ήθελα να σας θέσω μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση για ένα project με το οποίο ασχολείται η ΕΖΑ και που γίνεται στη χώρα μου, στις, στην Σαζόρες. Ήθελα να γνωρίζω λοιπόν ποια είναι η γνώμη σας, ε, να δούμε ποια Ποια είναι η θέση αυτού του project μέσα στη Γενική Στρατηγική 4.0. Η ΕΖΑ μαζί με την ΆΖΑ και με την Βραζιλιάνικη Διαστημική Υπηρεσία έχουν φτιάξει την πρωτοβουλία του ΕΡΑ ε, ε, Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο των Αζωρών ε, για οι Αζόρες πάντοτε ήταν μια βάση γεωστρατηγική πολύ σημαντική στο πλαίσιο όλων των μεγάλων συγκρούσεων ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα έχει μετατραπεί σε μια βάση στο πλαίσιο της ειρήνης που θέλουμε να επικρατεί στον κόσμο και μέσα εκεί περιλαμβάνεται ε, η βάση εκτόξευσης χαμηλού κόστου ε, υπάρχουν συγκεκριμένα οχήματα, έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την στρατηγική για την μάλλον γεωεντοπισμό ε, από πλευρά τη ΝΑΖΑ. Έχουμε συνεργασία με την Ισπανία, τη Βραζιλία, ε, χώρε τη Λατινική Αμερική και τη Αφρική, ε, τη ΣΥΠΑ και ούτω καθεξή. Θα ήθελα να μα πείτε κάποια πράγματα περισσότερο όσον αφορά τη σημασία που αποδίδεται σε αυτό το project μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μούντι. Σας ευχαριστώ πολύ. Your inspiring presentation. Και σας ευχαριστώ για την πολύ εμπνευσμένη σας ε, ομιλία. Ως Βρετανίδα δεν θα σας εντυπωσιάσει που μου άρεσε ιδιαίτερα εκείνη η slide, εκείνη η διαφάνεια με τον Team Peak και το γαλλικό κανάλι. Ναι, σίγουρα μας χρειάζεται λίγο περισσότερο ευρωπαϊκό πνεύμα ε, στην χώρα μου. Ε, εν πάση περιπτώσει πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικό τομέα ε, όπου καλύπτει ζωτικά στοιχεία ε, και φυσικά είναι πολύ σημαντικό ότι προσφέρεται θεμελιώδη στήριξη. Έχουμε στην περιφέρειά μου το Μεταλφής και ξέρω πάρα πολύ καλά ποια είναι τα ωφέλη που προκύπτουν από την διαστημική μας πολιτική. Τώρα, ε, όσον αφορά τη βιομηχανική πολιτική, και εδώ συνδέουμε με κάτι που ήδη έχει υποθεί, έχουμε τη σημασία των μικρών δορυφόρων και τον όγκο καινοτομία που μπορεί να ε, υπάρξει μέσω των μικρών δορυφόρων. Εκεί θα ήθελα κάποια περισσότερη σαφήνεια και για το πώς εκτοξεύονται. Πράγμα που με φέρνει και σε κάτι το οποίο δροθυγώς αναφέρατε στην εισήγησή σας, αλλά θα ήθελα κάποια μεγαλύτερη ε, ανάπτυξη. Τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες για την τεχνολογία οριζόντιας εκτόξευσης. Ε, ε, Πάντως, ε, οι τρεις λέξεις που για μένα με, μου έμειναν είναι η περιέργεια, έπνευση και συμμετοχή ε, στη δική σας εισήγηση. Και πιστεύω πως χρειάζεται να υπάρχει περισσότερη στήριξη για αυτό το στοιχείο της περιέργειας από ό,τι βλέπουμε στην ίδια τη στρατηγική και στο σχετικό, στη σχετική ανακοίνωση μέχρι τώρα. Μιλήσατε ότι από με βάση αυτή τη τεχνολογία πυροδοτούνται και άλλες εξελίξεις. Έχουμε, υπάρχουν ένα σωρό σχολεία που ασχολήθηκαν με τον Τιμ Πίκ όταν ε, πήγε στο διάστημα και πραγματικά η νέα γενιά αρχίζει να καταλαβαίνει τον τομέα του διαστήματος χάρη σε αυτή την υπόθεση και πολλά συζητήθηκαν. Συζητήθηκαν, ε, είπαμε, ας πούμε, πώς βλέπουμε τον εαυτό μας από το διάστημα ε, αλλά και πώς μπορούμε πέρα από τον εαυτό μας να κοιτάξουμε μέσα στο διάστημα ε, ε, και αυτό έχει να κάνει με την περιέργεια, την έμπνευση και τη συμμετοχή γιατί εκεί μπορούμε να δείξουμε ότι προστιθέμενη αξία δίνουμε κάτι το οποίο δεν υποκαθιστά τα όσα κάνουμε για να επεκτείνουμε και να διανοίξουμε τους ορίζοντές μας. Ευχαριστώ συνάδελφε. Να προσθέσω Κύριε Γενικέ Διευθυντά, σίγουρα είστε ε, παδός της ε, διαστημικής πολιτικής αλλά και της ε, ολοκλήρωσης ε, μ' αρέσει να δίπλα-δίπλα αυτές οι λέξεις. Είπατε για κάτι το πολύ γοητευτικό και πολύ σημαντικό από την άποψη της ολοκλήρωσης. Ε, ε, γιατί ε, εξάλλου μπορεί κανείς να τα βρει όλα στο ίντερνετ και οι νέοι μπορούν να τα βρουν όλα στο ίντερνετ δεν χρειάζεται να τους διδάξουμε αλλά μπορούμε να τους δώσουμε προτάσεις για 2, 3, 4, 5 μαθήματα θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα Διαστημική πολιτική και ολοκλήρωση. Τι λέτε. Και έτσι ολοκληρώνεται η, συνεδρία των ερωτήσεων. Περνάμε στη συνεδρία των απαντήσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τα καλά σας λόγια. Τα δέχομαι. Είναι καλό να ακούει καλές πένους, σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα. Τώρα, κάποιες ερωτήσεις συνδέονται μεταξύ τους. Αν μου επιτρέπετε, θα τα πω κάπως πιο συμπυκνωμένα. Θα απαντήσω πιο ομαδικά. Έζα και... Ε, ε, ποια είναι τα project τα που κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να μην είμαστε ανταγωνιστές. Θα πρέπει να είμαστε συντονισμένοι και να συνεργαζόμαστε. Υπάρχει ένα μέσο στην Διοργανική Συμφωνία που αναφέρεται το 2004 ανάμεσα στην ΟΗΕ και την ΒΕΖΑ ότι θα που λέει ότι πρέπει να υπάρχει ε, μια ε, διαστημική συνεργασία. Είναι άτυπες όμως σκέψεις που βασίζονται σε μια τυπική ε, συμφωνία πλαίσιο. Δεν θα πρέπει νομίζω να βλέπουμε εμεί τώρα ποια νομική κατάσταση, θα πρέπει να συνεδριάζουμε η ΕΖΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δούμε τι είναι καλό για το μέλλον όλων μας και σε αυτό να προχωράμε. Και βέβαια έχουμε διάφορες αρμοδιότητες και πρέπει να τις χρησιμοποιούμε. Η Κομισιόν έχει ισχυρή αρμοδιότητα στις τομεακές πολιτικές. Και αυτό επανέρχεται σε μια ερώτηση. Χρήση του διαστήματος για τη γεωργία ή για την αυσιπλοεία ή για την ε, ρύθμιση της κυκλοφορίας και ούτω καθεξής. Οι τομεακές πολιτικές είναι η ισχύση της Επιτροπής, ενώ εμείς στην ΕΖΑ ξέρουμε πώς να τα θέσουμε σε εφαρμογή. Έχουμε την τεχνολογία, την Αυτά λοιπόν μπορούν πολύ ωραία να συντεριαστούν γι' αυτό και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιοριζόμαστε σε ένα από αυτά τα projects. Θα πρέπει να διερευνούμε διάφορους δρόμους και να τους συνδυάζουμε. Γαλιλαίο και Κοπέρνικος είναι καλό παράδειγμα για το τι μπορούμε να καταφέρουμε. Και υπήρξε ένα θέμα για το πώς ε, ε, ξεκίνησε στο Γαλιλαίο η ιδέα ήταν να έχουμε 27 διαφορετικούς δορυφόρους σε διαφορετικές τροχιές γιατί ε, αν τους βάλεις όλους στην ίδια τροχιά δεν μπορείς να έχεις το ε, σήμα πλοήγησης. Και να έχουμε και τρεις εφεδρικούς ε, στο έδαφος. Αν οποιοδήποτε δηλαδή δορυφόρος χαλάσει, που μπορεί να συμβεί, να μπορείς να τον αντικαταστήσεις με έναν άλλον στην ίδια τροχιά. Νομίζω ότι το 2028 ε, θα έχουμε πλήρη, τον πλήρη αυτό αστερισμό. Τέσσερις έχουν ε, εκτοξευθεί, έχουμε ε, τον Αριά, την Αριάν. Ακούγεται εύκολο, αλλά πρέπει να φτάσουν σε διαφορετική τοποθεσία στο διάστημα. Πάει, μπαίνει στην τροχιά του το διαστημόπλιο, μετά απελευθερώνει δύο δορυφόρους και μετά απελευθερώνει άλλους δύο δορυφόρους. Πολύ τεχνικό ζήτημα. Ε, οι επιχειρήσει αυτές έγιναν και ευτυχώ είχαν αίσιο πέρας. Ε, Έχαμε και τον Τωμά Πεσκή που έπρεπε να εκτοξευθεί την περασμένη εβδομάδα και έναν Ευρωπαίο αστροναύτη με γαλλικό αξό. Ε, ε, ε, έχουμε πάρα πολύ αξιόπιστου εκτοξευτές. Έχουμε 75 εκτοξεύσεις επιτυχής στη σειρά, χωρίς αποτυχία. Είναι το ρεκόρ μας. Περισσότερο και από το Ιναριάν 4, αλλά ο ανταγωνισμό είναι πολύ ισχυρό και γι' αυτό πρέπει να έχουμε έναν πιο φτηνό εκτοξευτή για το μέλλον. Η Ιναριάν 6 θα είναι 50% φθηνότερη από την Ιναριάν 5 θα είναι έτοιμη το 2020 και ταυτόχρονα αναπτύσσουμε και το Vega 6, ένα μικρότερο εκτοξευτή, ώστε στο μέλλον θα έχουμε μια μεγάλη οικογένεια εκτοξευτών. Το μικρότερο είναι Vega 6, το μεγαλύτερο λίγο είναι η Ariane 62 που έχει δύο τουρμπι, ε, τουρμπίνες, όπως η μηχανή και του Vega 6 και μετά θα έχουμε την Αρένα 64 με 4 ε, ε, ε, τουρμπίνες. Έχουμε μια οικογένεια και αυτό κάνει και φθηνότερη την κατασκευή. Πολύ ελκυστικό μέλλον, λαμπρό μέλλον προβλέπεται. Έχουμε δηλαδή το, για το 23 προβλέπεται η ανάπτυξη και του Άρια 6 αλλά θέλουμε και τις ιδέες για τις νέες τεχνολογίες και βεβαίως επισκέφθηκα τους ε, κινητήρες και τις νέες ιδέες τις χρειαζόμαστε για το μέλλον, για τους εκτοξευτές και να μην κοιτάμε τους Αμερικανούς και να λέμε υπάρχει και ένας που χρησιμοποιεί το Tesla και τώρα ο Έλαν Μάσκ ε, κάνει ε, πολλαπλών χρήσεων εκτοξευτέ. Δεν ξέρω, αν δείτε εδώ αυτό το, το μπουκάλι, έχουμε διαφορετικών ειδών μπουκάλια. Έχουμε αυτά που είναι πολλαπλών χρήσεων, έχουμε τα ανακυκλώσιμα μπουκάλια και έχουμε και γυάλινα μπουκάλια. Ε, οπότε δεν έχουμε μια τεράστια αγορά. Εδώ έχουμε μικρό αριθμό ε, εκτοξευτών, δεν είναι αγορά ε, μάζας μεγάλη μάζα. Έχουμε έξι εκτοξεύσεις το χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια λύση οικονομική για μας, για εδώ, για την Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και πιο ριζοσπαστικέ τεχνολογίε. Επίση, σε δύο μέρες θα παρουσιάσουμε στα κατημέλη, σε δύο μέρες, μια ε, πρωτοβουλία για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 10 και για μικρού δορυφόρου, πολύ μικρού δορυφόρου. Και νομίζω πως ε, αυτή είναι πολύ καλή ιδέα γιατί συνδέεται και με τις ανάγκες της βιομηχανίας που αναφέρατε. Φυσικά και ε, όπως σας είπα ο ανταγωνισμός είναι διαφορετικός στην Ευρώπη από ότι στην ε, ΣΥΠΑ έχουμε ομίλου αλλά και μικρομεσαίε επιχειρήσει και στην ΕΖΑ έχουμε ειδικό πρόγραμμα για να τις στηρίξουμε, για να τι φέρουμε σε επαφή με τα στοιχεία μα, γιατί ζητούσατε για την πολιτική, ρωτήσατε για την πολιτική στοιχείων. Έχουμε μια πολιτική ελεύθερων δεδομένων. Δεν ήταν ε, τόσο εύκολο να πείσουμε του δικού μα ότι ήταν αυτή η καλή λύση, αλλά υπάρχει. Για το κοπέρνικο, α πούμε, για την παρατήρηση τη γη, είναι ανοιχτά. Αλλά ανοίγουμε και όλα μα τα βιβλία για τα τεχνικά στοιχεία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα και για τα επιστημονικά στοιχεία. Στον επιστημονικό τομέα έχουμε περίπου έξι μήνες καθυστέρηση. Θα είμαι πολύ ε, ε, ειλικρινής, γιατί ο κύριος ερευνητής θα ήθελε να έχει το δικαίωμα της πρώτης ε, της παρουσίασης των στοιχείων του της πρεμιέρας και για τα επιστημονικά στοιχεία έχουμε έξι μήνες καθυστέρηση μέχρι ότου να ε, ε, δημοσιευτούν τα στοιχεία. Και γι' αυτό δεν είμαστε μόνο χρηματοδότης, αλλά αποτελούμε και μια βάση διευκόλυνσης για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και του κλάδου αυτού. Αυτά. Και μετά, για την παιδεία. Εγώ ελπίζω. Η απόδοση επί των επενδύσεων είναι θετική, αλλά η απόδοση επί των επενδύσεων δεν σημαίνει χαλάω ένα ευρώ ή μια λίρα σήμερα και αύριο παίρνω πίσω έξι γιατί αυτό είναι περίπου η αναλογία στη, για το διάστημα. Ε, η απόδοση είναι ένα, ο λόγος είναι ένα προ έξι όσον αφορά την απόδοση. Κάποιε φορές πρέπει να περιμένουμε περισσότερο για την απόδοση και να έχουμε διαφορετικού είδους απόδοση. Αν πρόκειται για έμπνευση, έμπνευση, γοητεία, κίνητρο για τη δημιουργία του μέλλοντος. Δεν είναι μόνο νέα τεχνολογία, δίνει, προσφέρει στον κόσμο ένα όνειρο. Η μητέρα μου, εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου είχαν όνειρα για μένα και μου μετέδωσαν αυτήν την προσδοκία να κάνω κάτι καλύτερα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Όλμπερτ Άινστάιν πριν από 100 χρονιά έγραψε τη θεωρία της σχετικότητας. Εντάξει, ξέρετε τις λεπτομέρειες όλοι. Υπάρχει ειδική θεωρία και η γενική. Η μία θεωρία λέει ότι ο χρόνος, ο χρόνος που βλέπουμε στο ρολόι μας εξαρτάται από τη βαρύτητα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά το πιστεύω και ο χρόνος εξαρτάται και από την ταχύτητα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Το προσπάθησα με το αυτοκίνητό μου, δεν είδα καμία διαφορά. Τώρα με τον Γαλιλαίο έχουμε σε τροχιά δορυφόρους που είναι πάρα πολύ γρήγοροι, ταχύς. Οπότε ο χρόνος αλλάζει γιατί οι δορυφόροι είναι τόσο γρήγοροι και υπάρχει ένα ρολόι πάνω στο, στους δορυφόρους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το δορυφορικό σύστημα πλάγησης. Ο χρόνος αλλάζει γιατί αυτοί οι δορυφόροι είναι τόσο γρήγοροι. Έπειτα, ο δορυφόρος ε, βρίσκεται σε ε, μια περιοχή με μικρότερη βαρύτητα. Άρα πάλι αλλάζει ο χρόνος εκεί. Αν δεν ξέραμε τα όσα είπε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν τότε, τα ασφάλματα θα ήταν 500 μέτρα σε μια ώρα για την πλοήγηση. 100 χρόνια Λεφτά δεν έχει, όμως έχει έμπνευση, επιστημονική έμπνευση και ξαφνικά ανοίγει ένας ολόκληρος νέος κόσμος μπροστά μας. Παιδεία λοιπόν, παιδεία και συμφωνώ μαζί σας ότι ε, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι σημαντικό. Και να σας πω για ακόμα τρεις ώρες αν με ξανακαλέσετε τι κάνουμε, έχουμε εκπαιδευτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα φυσικά και θέλουμε περισσότερη στήριξη γι' αυτό. και θα πρέπει να δοθούν και υποτρεφίες σε φοιτητές, σε σπουδαστές, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, ε, τα απόβλητα του διαστήματος, τα σκουπίδια του διαστήματος υπάρχουν για το μέλλον, δεν είναι επικίνδυνο και ξέρω κανείς δεν θέλει να το, δεν θα το καταλάβει, θέλω να πω ένα αλλά κανείς δεν το καταλαβαίνει. Χρειαζόμαστε μια ηλεκτρική σκούπα του διαστήματο να καθαρίσει το κενό. Ναι, ειδικά οι Βρετανοί θα πούνε ναι, σκούπα ηλεκτρική έχουμε σπίτια μας. Ε, χρειαζόμαστε εδώ όμω έναν καθαριστή του κενού στην ουσία, vacuum στα αγγλικά. Ε, είναι δύσκολο όμω να το εκτιμήσουμε και πώς θα λειτουργήσει. Το ίδιο γίνεται και όταν αγοράζεις ένα νέο προϊόν. Πληρώνεις πολλά, αν θες να το ξεφορτωθείς δεν πληρώνεις τα ίδια γιατί ε, αγοράζεις κάτι καινούριο και απλώς το πετάς μια ηλεκτρική σκούπα για το κενό λοιπόν θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ίσως και σε παγκόσμιο. Τώρα, η πλανητική αμήνα τώρα είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, να είμαστε βέβαιοι ότι ένας, ένας μετεωρίτης ή, οτιδήποτε άλλο ε, πέφτει πάνω μας να μπορούμε να αμυνθούμε. Δεν είναι στρατιωτικό, πρόκειται για προστασία του πολίτη, αλλά είναι άμυνα. Πλανητική άμυνα και μετά έχουμε και την πλανητική προστασία. Γι' αυτό επανέρχεται στα ερωτήματά σας. Ε, να μην ρηπαίνουμε άλλους πλανήτες. Υπάρχει η ιστορία του Απόλλω 12 ε, που προσιώθηκε στη Σελήνη και πήγε σε ένα μικρό ε, διαστημόπλαιο νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήτανε, το άλλο διαστημόπλαιο και βγάλαν το κάμερα από εκείνο το ρομποτικό διαστημόπλαιο, την έφεραν στην, στην γη και ασχολήθηκαν μαζί του και βρήκαν κάποια βακτήρια. Και βέβαια ήταν πολύ περίεργεια ότι ζούσαν βακτήρια στο φεγγάρι. Όχι, ήταν ο τεχνικός που κατασκεύασε την κάμερα που ήταν κρυωμένος. Και τα προσπαθούμε λοιπόν να τα ερευνήσουμε. Όλα αυτά τα, τα προϊόντα πρέπει να είναι πολύ καθαρά ώστε να μην μολύνουμε το σύμπαν μας. Τελευταία ερώτηση. Να σας πω, χρειάζεται και στο μέλλον η δυνατότητα να ερευνήσουμε ε, σε περιβάλλον ε, μικροβαρύτητας ή ουδέτερης βαρύτητας. Γιατί η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί στο διάστημα. Έχουμε νέα βιολογικά πειράματα με ανθρώπους όμως πρέπει να γίνουν. Αν δεν βάλουμε τους ανθρώπους στην μικροβαρύτητα, χάνουμε την ευκαιρία να ερευνήσουμε την, ε, ε, ε, τη δυνατότητα. Αλλάζουν όλα. Αλλάζουν όλα, ας πούμε, για την οστεοπόρωση και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις υποσημονικές έρευνες και οι επιστήμονες είναι ευτυχείς μόλις βρουν ένα δίκτυο και τον αλλάξουν και κάτι άλλο γίνεται. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για ιατρικά προϊόντα, ήδη χρησιμοποιείται για την οστεοπόρωση κυρίως Πρέπει να καταστεί δυνατή η έρευνα στη μικροβαρύτητα και μετά από το ISS, θα πρέπει, το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, θα πρέπει να φτιάξουμε ένα νέο, θα πρέπει να φτιάξουμε νέες παγκόσμιες έρευνες και μετά φτάνουμε και στα ε, φεγγαροχωριά, ε, τα χωριά στο φεγγάρι, δεν είναι project, είναι μια ιδέα, είναι μια ανοιχτή ιδέα, σαν να είναι να φτιάξουμε ένα χωριό στην γη. Και ελπίζουμε πως έτσι θα δώσουμε έμπνευση και ε, διεθνή συνεργασία. Ελπίζω πως πάνω κάτω απάντησα στα όσα μου ρωτήσατε, αλλά ε, ε, μπορώ να πω κι άλλα, αλλά υπάρχουν και περιορισμοί. Ναι, ξεχάσα τις Αζόρες, συγγνώμη, στις Αζόρες υπάρχει μια δραστηριότητα τα τρία α, Ακτική, Ατλαντικό και η άλπις. Τι σχέση έχουν αυτά τα τρία θα μου πείτε το συζητήσαμε και χρησιμοποιούμε ε, για θαλάσσιες δραστηριότητε πλέον και εφαρμογές ε, από το διάστημα. Η Αρκτική αφορά, όπως ξέρετε, τις χώρες χώρες και οι Άλπες είναι σαφές, καταλαβαίνετε. Ναι, Έχουμε ακούσει όλοι για τη θεωρία του Einstein, αλλά δεν την καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά, δυστυχώ. Λοιπόν, αυτό το, το χωριό στο φεγγάρι, ε... είχα μια συνάντηση με 800 ανθρώπους περίπου, έγινε παρουσίαση για τη στρατηγική για το διάστημα και έγινε αναφορά σχετική με εξαιρετική ιδέα τώρα. Ε, δεν ξέρω καθόλου τι είναι όμως. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Καλή ιδέα πάντως φαντάζομαι. Αγαπητοί φίλοι, ήταν η πρώτη συνάντηση. Ελπίζω να δούμε συχνά τον Διευθυντή, τον κύριο Βέρνερ, στα επόμενα δυόμιση έτη της θητείας μας στην Επιτροπή αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σας και για τον ενθουσιασμό σας. Είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενθουσιασμός. Ε, dear friends. Αγαπητοί φίλοι, θα ξαναξαναπούμε εδώ στις 3 ακρόαση για το μέλλον της έρευνας στην Ευρώπη.